Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε. Ναι. Ξέρω ότι σήμερα είναι Δευτέρα. Μάλιστα έχουμε και ένα τραγούδι στα πολωνικά, δεν μου αρέσουν οι Δευτέρες. Αλλά παρόλα αυτά θα ήθελα να ξεκινήσουμε. Σας καλωσορίζω θερμότατα στη συνεδρίασή μας. Έχουμε μια κοινή ακρόαση σήμερα με την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Έχουμε κάποιες κοινέ αρμοδιότητες με την Επιτροπή ΕΜΒΗ για τα θέματα ασφάλειας των τροφίμων είναι συνδεδεμένες οι δύο Επιτροπές, Γεωργίας και Περιβάλλοντος. Δεν θα ήθελα να περάσω ακόμη στο επίσημο ε, τμήμα της ακρόασης που θα γίνει με συμπροεδρία των δύο ε, επιτροπών. Θα έρθει σε λίγο η κυρία Βαλεάν που είναι η πρόεδρος Επιτροπής ΕΜΒΗ και θα προεδρεύσει το δεύτερο πάνελ τη ακρόαση. Να σα ενημερώσω ότι η ερμηνεία υπάρχει σε 20 γλώσσε με εξαίρεση τσεχικά, μαλτέζικα, σλοβακικά και κελτικά, ιρλανδικά. Και να καλωσορίσω εκ μέρου τη Επιτροπή μα του ευρωβουλευτέ και του καλεσμένου στη δημόσια ακρόαση με τίτλο «Η επισήμανση τη προέλευση στα γεωργικά προϊόντα και τα προϊόντα διατροφή. Επαναλαμβάνω, πρόκειται για κοινή ακρόαση δύο επιτροπών. Ε, θα ήθελα να πω ότι στην συζήτηση, στην ακρόαση αυτή θα εξετάσουμε κυρίως την εφαρμογή των εθνικών συστημάτων επίσημα στα κράτη-μέλη και θα εξετάσουμε από εκείνο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον εκτελεστικό κανονισμό ε, και κυρίως ε, την εθελοντική αναφορά της χώρας καταγωγής ή τόπου προέλευσης για τα τρόφιμα βάσει το άρθρο 23.3 του κανονισμού 1169 του 201 που πρόσφατα εγκρίθηκε και θα δούμε κατά πόσο είναι ε, επαρκής ανταπόκριση στα αιτήματα των καταναλωτών για περισσότερη διαφάνεια. Γιατί οι καταναλωτές φαίνεται ότι ζητούν επίμονα την αναφορά της ε, χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης από τα τρόφιμα χάρη μεγαλύτερης διαφάνειας. Θα ήθελα να καλωσορίσω τώρα την κυρία Αντίνα Γιώνα Βαλεάν, την πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που θα συμπροεδρεύσει μαζί μου σε αυτή τη δημόσια κρόση. Και να ευχαριστήσω θερμά και τον κύριο Καπούτο, αλλά και όσους συνέβαλαν στη διοργάνωση της σημερινής ακρόασης. Ελπίζω ε, να καταφέρουμε χάρη στην ακρόαση να διαμορφώσουμε μια πιο γενική αντίληψη και πιο εμπεριστατωμένη της εμπειρίας και των αποτελεσμάτων που επέφερα στα κράτη-μέλη τα εθνικά συστήματα εφαρμογής και να δούμε πώς ε, αξιολογείται ο αντίκτυπος αυτών των συστημάτων σε ενδιαφερόμενους στο κλάδου όπως στην αλυσίδα τροφίμων κυρίως και στους γεωργούς θα ακούσουμε στη διάρκεια της ακρόασης ε, μερικές εθνικές εμπειρίες στο πρώτο πάρελ και στο δεύτερο πάρελ θα πρέπει να απαντήσουμε στην ερώτηση αν ο εκτελεστικός κανονισμός ε, ε, που προβλέπει την επισήμαση της, στην, στο τρόφιμο της χώρας καταγωγής της, του τόπου προέλευσης είναι ε, επαρκής απάντηση στην απέτηση των καταναλωτών για μεγαλύτερη διαφάνεια και ανταποκρίνεται επίση ανάγκε ε, των ε, διαφόρων παραγόντων τη τροφική αλυσίδα και κυρίω των γεωργών. Σε αυτό το ερώτημα θα κληθούμε να απαντήσουμε στο δεύτερο πάνελ. Και να καλωσορίσω του εμπειρογνώμονέ μα. Ε, θα μιλήσουν και θα ακολουθήσει συζήτηση με ερώτα απαντήσεις. Ε, στο δεύτερο είπα, τμήμα της δημόσιας ακρόασης θα προεδρεύσει η πρόεδρος της ΕΒΗ κυρία Βαλέαν και θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε άλλους τρεις καλεσμένους και εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας. Επίσης, να τονίσω ότι έχουμε πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα και είναι σημαντικό να τηρήσουμε το χρόνο αγόρευση. Θα ακούσουμε στο πρώτο πάνελ κάποιες εθνικές εμπειρίες κατά την εφαρμογή των εθνικών συστημάτων. Ο πρώτος καλεσμένος μας είναι ο κύριος Ρομπέρτο Μονκάλβο, πρόεδρος ε, της ε, Ιταλικής Ένωσης του Ιταλικού Συλλόγου Γεωργών Κολντιρέτη. Θα μας παρουσιάσει την Ιταλική εμπειρία. Κατόπιν ο κύριος Σεμπάστια Χίλμα, που είναι Διευθυντής Ασφάλειας Τροφίμων στο Φιλανδικό Υπουργείο Γεωργίας και δασοκομείας θα μας παρουσιάσει την εμπειρία της Φιλανδίας και η κυρία Καμίχ Πέρα που είναι αρμόδια σε θέματα πολιτικής τροφίμων από την Ευρωπαϊκή ε, Οργάνωση Καταναλωτών θα μας κάνει μια γενική παρουσίαση και κατόπιν θα μας αναφέρει την εμπειρία της Γαλλίας. Παρακαλώ 10 λεπτά ο καθένας και πρώτος έχει το λόγο ο κύριος Μονκάλβο στον οποίο και δίνω το λόγο. Παρακαλώ 10 λεπτά και όχι παραπάνω. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δώσατε το λόγο. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Ρομπέρτο Μονκάλβο, προεδρεύω της Κολτιρέτη, είμαι 37 ετών, Γιώργος. Η Κολτιρέτη έχει 1,6 εκατομμύρια μέλη στην Ιταλία και είναι η πιο μεγάλη ένωση της κατηγορίας αυτής στην Ιταλία και συνεργάζεται με διάφορους φορείς που προωθούνται από την Κολτιρέτη και επεξεργάζεται βασικά θέματα της, των τροφίμων και της γεωργίας στην πατρίδα μου. Βλέπετε στην πρώτη διαφάνεια είναι η Fondazione Καμπάνα Μίκα, είναι μια ένωση στην οποία έχουμε εκατομμύρια μέλη, Ιταλούς πολίτες, που διοργανώνουν αγορές ε, ε, των ε, διαφόρων αγροκτημάτων και κάνουν απευθείας πωλήσει διαφόρων ε, προϊόντων και έχουμε 1.200 αγορές που οργανώνουμε και συμμετέχουν ε, περίπου 20.000 εκμεταλλεύσεις. Έχουμε το παρατηρητήριο της, ε, των απατών. Βλέπετε ότι οι βασικοί εισαγγελείς συμμετέχουν, οι δυνάμεις του τάξη συνεργάζονται με την Κολτιρέτη για να δημιουργήσουν, θεσπίσουν νέα νομοθεσία και κανόνες για να καταπολεμήσουν την απάτη στον τομέα των αγροτριφημικών. Έχουμε την Credit Agri, είναι ένα consortium εγγύησης ε, που παρέχει εγγύσεις για επενδύσεις στις ε, αγροτικές εκμεταλλεύσεις ε, και χρηματοδοτεί πάνω από 4 δις ευρώ. Και έχουμε τη Φιλιά Ρετάλια, μια ένωση στην οποία η Γεωργία Βιομηχανία και οι διαφασικές βιομηχανίες της χώρας και οι κοντιρέτοι συναντώνται και συνομιλούν και συζητούν αυτά τα θέματα που αφορούν την ετικεταθεσία και την προάσπιση των Ιταλικών και Ευρωπαϊκών τροφίμων. Γιατί είναι σημαντική περισσότερη διαφάνεια και περισσότερες πληροφορίες που χορηγούνται στους καταναλωτές. Να σας πω τι λέει το Υπουργείο Γεωργίας της Ιταλίας. Με δημοσκοπήσεις επίσημες απέδειξε αυτό που λέμε επί σειρά ετών στην Κοντιρέτη. Ότι 96% των Ιταλών πολιτών ζητούν υποχρεωτικά να αναφέρεται η προέλευση στην ετικέτα των τροφίμων. Και 80% των Ιταλών πολιτών θεωρούν σημαντικό να αγοράζουν τρόφιμα made in Italy που παράγονται με γεωργικά συστατικά που είναι, έχουν παραχθεί στην Ιταλία. Αυτό ε, είναι πολύ σημαντικό θέμα και τους πρώτους μήνες του 2018 ακόμα δηλαδή μετά τη δημοσίευση της εκτελεστικής πράξης του κανονισμού 1169 ε, ε, έγινε επίσης μια κινητοποίηση των πολιτών που ζητούν υποχρεωτική αναφορά ε, των πληροφοριών και συλλέξαμε πάνω από 200.000 υπογραφές σε δύο μήνες για αυτή την υποχρεωτική επισήμανση. Ποια είναι η αξία αυτού. Ε, ανταποκρίνεται στην απέτηση των πολιτών για διαφάνεια και μετά μας επιτρέπει αυτό να είναι αναγνωρίσιμη η δουλειά των γεωργών μας σε σχέση με την βιωσιμότητα και την ποιότητα της παραγωγής και μπορούμε βέβαια και να εργαστούμε το ώστε να αποφύγουμε το φαινόμενο του sounding που δεν είναι μόνο ε, ιταλικό αλλά όλες τις χώρες που έχουν ε, που γίνεται αντιγραφή των προϊόντων από τίτες χώρες φαινόμενο αντίχηση στο Λοιπόν, την πρώτη εμπειρία που είδαμε μετά την εφαρμογή του νόμου της, του διατάγματος αυτού του εθνικού που εφαρμόζεται εδώ και πάνω από ένα χρόνο αφορά το γάλα και τα παράγωγα του γάλακτος ε, αυτή η επισήμανση. Το διάταγμα αυτό λοιπόν, το Ιταλικό, προβλέπει τον, την αναφορά της χώρας ε, που έγινε το άρμεγμα και εκεί που έγινε η μεταποίηση του τελικού προϊόντου. Μπορεί να είναι ένα γιαούρτι, μπορεί να είναι ένα τυρί ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν γάλακτος, το τελικό προϊόν. Με το ίδιο σχήμα, πρόγραμμα όπως αφορά το γάλα και τα τυριά και τα άλλα γαλακτοκομικά, κατόπιν ετήματος της Κολντιρέτη, επίσης έχουν βγει διατάγματα για υποχρεωτική αναφορά προέλευσης και για την παραγωγή επίσης του σκληρού σιτού, για την παραγωγή των μακαρονιού, ε, του ε, ρυζιού και των παραγόγων της ντομάτας. Ε, βλέπετε εδώ κάποια παραδείγματα ετικετών που στην Ιταλία πλέον βρίσκονται στο εμπόριο, στα προϊόντα, εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο. Μπορούμε να ξεκινήσουμε να αναλύουμε και τις θετικές συνέπειες της υποχρετικής αναφοράς προέλευσης στην ετικέτα, σε αυτή την περίπτωση για το γάλα και τα προϊόντα γάλακτος. Τον τελευταίο χρόνο, παίρνοντας τα επίσημα στοιχεία Νίλσεν όσον αφορά τη τιμή του γάλακτος στην κατανάλωση, τι είδαμε, ότι η τιμή του γάλακτος ουσιαστικά παρέμεινε σταθερή. Αυξήθηκε σε ένα χρόνο κατά 0,6%. Σχεδόν αμετάβλητη τιμή του γάλακτος. Αυτό που άλλαξε πολύ όμως είναι η τιμή που, που πληρώνεται για το γάλα στους φινοτρόφους μας. Η αναγνωρισμένη τιμή του γάλακτος αυξήθηκε τους τελευταίους 18 μήνες τουλάχιστον κατά 25% αυτό που καταβάλλεται στους ε, κτηνοτρόφους. Οπότε αυτό μας οδηγεί στο να πούμε ότι έχουμε δώσει απάντηση σε απαιτήσει των καταναλωτών που ήθελαν να έχουν υποχρετική αναφορά προέλευση στο γάλα και, και, και αναφορά γίνεται και στο τυρί δεν επιδεινώσαμε, δεν αυξήσαμε το κόστος αγοράς γάλακτος και παραγόγων γάλακτος για τους πολίτες καταναλωτές γιατί η τιμή παρέμενε ουσιαστικά αμετάβλητη αλλά έγινε μια ανακατανομή της αξίας σε όλη την αλυσίδα παραγωγής και τελικά ωφελήθηκαν οι ε, κτηνοτρόφοι που είδαν η τιμή του γάλακτος, η τιμή του γάλακτος στην εκμετάλλευση να αυξάνεται κατά 25% το τελευταίο 18 μήνο. Όπως σας έλεγα, αυτή η εμπειρία από το γάλα πρόσφατα επαναλήφθηκε αυτό το πείραμα και είμαστε στα πρώτα, στους πρώτους μήνες εφαρμογής και στο σκληρό σύτο για τα ζυμαρικά, για το ρύζι και για τα παράγωγα της ντομάτας. Οπότε παρακολουθούμε καθημερινά την κατάσταση για να αξιολογήσουμε τις συνέπειες που θα έχουμε στο εγγύς μέλλον. Και έχουμε άλλες 7 ευρωπαϊκές χώρες που έκαναν πειράματα ανάλογα με αυτά της ε, Ιταλίας μέσω εθνικών διαταγμάτων για την υποχρεωτική ετικετοθεσία που αφορά την παραγωγή των προϊόντων. Είναι προφανές ότι κατά την άποψή μας σήμερα το πρόβλημα είναι η έλλειψη εναρμονισμένων κανόνων στην Ευρώπη. Αυτή η έλλειψη κανόνων εναρμονισμένων στην Ευρώπη δεν μας επιτρέπει να ανταποκριθούμε στο αίτημα των πολιτών, δηλαδή υποχρεωτική αναφορά προέλευσης στην ετικέτα, αλλά πάνω απ' όλα δεν ε, ανταποκρίνεται επίση σε αυτό που το Ευρωκοινοβούλιο ε, και εσείς το σε αυτό επανειλημμένα ήδη έχει διακηρύξει σε τρία διαφορετικά ψηφίσματα στην τελευταία θητεία εσείς οι Ευρωβουλευτές του Ευρωκοινοβούλιο ε, δηλώσατε με μεγάλη πλειοψηφία ότι είσαστε υπέρ της υποχρετικής αναφοράς της προέλευσης του προϊόντος στην ετικέτα. Εάν δούμε τι συνέβη όμως με την έγκριση του κανονισμού του εφαρμοστικού τους πρώτους μήνες του 2018 βλέπουμε ότι αυτός ο εφαρμοστικός κανονισμός ε, στην πράξη δεν ανταποκρίνεται ούτε στις απαιτήσει των πολιτών καταναλωτών που ζητούν την υποχρεωτική αναφορά προελεύσεως στην ετικέτα του γεωργικού προϊόντου και των βασικών συστατικών σε κάθε τρόφιμο ούτε στις πολυάριθμες εκκλήσεις του Ευρωκοινοβουλίου ανταποκρίνεται η κατάσταση και στην πράξη σε πολλές περιπτώσεις συγχέεται η προέλευση του βασικού συστατικού με την τελωνιακή προέλευση των προϊόντων. Για μία ακόμη φορά ε, έγινε ένα μικρό βήμα πρόοδου, αλλά είναι θελοντικό το σύστημα και η προσέγγιση δεν είναι υποχρεωτική για όλους να αναφέρεται η προέλευση του προϊόντος στην ετικέτα. Και η παρέκκληση όσον αφορά τη γεωγραφική αναφορά και πάνω απ' όλα για τα εμπορικά σήματα είναι μια παρέκκληση η οποία επιδεινώνει περαιτέρω την εφαρμογή, τα αποτελέσματα του εφαρμοστικού κανονισμού και κατά την άποψή μας μάλιστα καθιστά αυτή την πράξη ε, ότι αντίθετα με αυτά που βλέπει το 26.3 του 1169 ε, του κανονισμού 1169 η παρέκκληση είναι πολύ πιο ευρία από ό,τι προβλέπεται. Να πω ότι αυτός ο κανονισμός, ο εφαρμοστικός, δεν λειτουργεί ως έχει και πιστεύουμε ότι είναι και, καινή ώρα πολιτικός να αντιμετωπιστεί το θέμα. Δεν ξέρω τώρα σε αυτή τη θητεία, στην επόμενη θητεία θα πρέπει να αλλάξει η κατάσταση, να αλλάξει ο κανονισμός ο βασικός ο 1169 για ούτω ώστε άπαξ απαντό για όλου του τομεί να υπάρχει υποχρέωση αναφορά προέλευση του ε, προβασικού συστατικού κάθε πρώτο τροφίμου και να ισχύει σε όλη την Ευρώπη και έτσι θα μπορούμε να ε, χρησιμοποιήσουμε όλα τα εθνικά, εθνικές προσπάθειες που γίνονται τους τελευταίους μήνες ξεκινώντας από την Ιταλία, από τη χώρα μου. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε και τώρα το λόγο έχει ο κύριος ε, Χέλμ από τη Φιλανδία. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι εδώ ε, στην Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να συναντώ τους ε, ευρωβουλευτές που είναι μέλη αυτής της Επιτροπής και άλλους που ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό. Σπάνια ε, ερχόμαστε σε επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συνήθως συζητάμε τα προβλήματα με την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δυστυχώς πολύ συχνά έχουμε διέξοδο. Καλύτερα να ερχόμαστε σε επαφή πιο συχνά με το Κοινοβούλιο για να μας βοηθήσει να ξεφύγουμε από αυτό το διέξοδο, γιατί αυτό το πρόβλημα έχουμε με την ε, με το θέμα της επισήμασης της προέλευσης. Θα σας παρουσιάσω ένα διάταγμα που έχει εκδώσει το Φιλανδικό Υπουργείο Γεωργίας και ε, δασοκομείας και ένα άλλο διάταγμα που δεν έτυχε θετική υποδοχής ε, επικρίθηκε από κάποιες χώρες και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε και αρνητική γνωμοδότηση για το δεύτερο αυτό φιλανδικό διάταγμα. Πάντως δεν έχει νόημα αυτή η αρνητική γνωμοδότηση. Εμείς θα συνεχίσουμε να τα εφαρμόζουμε για περιορισμένο χρόνο. Καταρχήν, να σας πω ότι το πρώτο διάταγμα είναι το 2017, της άνοιξης του 2017 και καθιστά υποχρεωτικό για τους παραγωγούς τροφίμων στη Φιλανδία να αναφέρουν στην ετικέτα την προέλευση κάποιων τροφίμων και του βασικού συστατικού τους. Μιλάμε για κρέας, που χρησιμοποιείται ίσω συστατικό σε προϊόντα διατροφή και μάλιστα χωρί ελάχιστο όριο. Αν ένα τρόφιμα περιέχει κρέα, θα πρέπει να αναφέρεται η χώρα προέλευση του κρέατος αυτού. Και υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να αναφέρεται η χώρα. Μπορεί να κατονομάζεται συγκεκριμένα η χώρα ή αν ε, το κρέας έρχεται από πολλέ χώρε μέλη θα μπορεί να αναφέρεται στην ετικέτα ότι είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή να είναι εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση ή EU ή non-EU. Άλλη ομάδα τροφίμων που καλύπτονται από το διάταγμα είναι τρόφιμα που περιέχουν ε, γάλα. Είτε κατανάλωση είτε ως ε, συστατικό για γαλακτοκομικά προϊόντα. Και μάλιστα δεν καλύπτονται όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα, αλλά μεγάλος αριθμός αυτό το προϊόντο που κανονικά έτσι τα αντιλαμβάνεται το κοινό. Και για αυτά τα προϊόντα τα γαλακτοκομικά περιέχουν γάλα, υπάρχει υποχρέωση αναφοράς της χώρας προέλευσης του γάλακτος. Τώρα, ερχόμαστε στο διάταγμα καθ' αυτό που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιουνίου του 2017 και θα κρατήσει μέχρι το Μάιο του επόμενου χρόνου. Διετές είναι αυτό το πιλωτικό διάταγμα. Εδώ έχει περιορισμένο πεδίο εφαρμογή, αφορά μόνο τα προσκευασμένα προϊόντα που, που παρασκευάζονται στη Φιλανδία και ε, ε, κατα... προορίζονται για την τελική κατανάλωση ή για τη μαζική εστίαση. Οπότε εδώ θα πρέπει να αναφέρεται η χώρα προέλευση για τα προϊόντα που περιέχουν κρέα ή γάλα, ενώ για, ξε... για εταιρείε που παράγουν τέτοια προϊόντα δεν καλύπτονται από αυτό το διάταγμα, αλλά θα ήταν αδύνατο να έχουμε ένα κανόνα που επεκτείνει αυτή την υποχρέωση και σε άλλες χώρες ε, προκειμένου να διαθέσει τα προϊόντα να υδαθέσουν τα προϊόντα τους στη Φιλανδία. Πάρος, πάντως παρόλα αυτά θεωρούμε ότι είναι πολύ αξιόλογο το διάταγμα και οι Φιλανδοί καταναλωτές ε, έμειναν ικανοποιημένοι από την εφαρμογή του και η παραγωγή μας το ίδιο και πιστεύουν ότι η εφαρμογή του διατάγματος αυτού θα είναι υποφελής ε, και για τους ίδιους, τους παραγωγούς. Τώρα, έχουμε και ένα σήμα χώρας προέλευσης ε, που ισχύει στη Φιλανδία εδώ και αρκετό καιρό. Είναι η ε, το σήμα που βλέπετε πάνω δεξιά στη διαφάνεια. Και ένας παραγωγός για να μπορεί να χρησιμοποιεί αυτό το σήμα, αυτή την ετικέτα στο προϊόν του, θα πρέπει να εγγυάται ότι η προέλευση ε, κρέατος, γάλακτος κρέατος πρέπει να είναι ε, σε μεγάλο βαθμό προ... φιλανδικό και το ίδιο και για τα προϊόντα. Ένα μεγάλο ποστό τους θα πρέπει να είναι ε, φιλανδικό. Και αν για κάποιο λόγο ένας παραγωγός ε, δεν θέλει να χρησιμοποιήσει αυτή την ετικέτα με τον κύκνο, θα πρέπει να αναφέρει τη χώρα προέλευσης, αλλιώς δεν χρειάζεται. Τώρα, δεν έχω συγκεκριμένε πληροφορίε αντίστοιχε με αυτέ του Ιταλού. Ξέρουμε ότι ήταν δημοφιλή αυτή την πρωτοβουλία και στου καταναλωτέ και στου παραγωγού και σε κάποιε εταιρείε παραγωγή τροφίμων, αλλά δεν έχουμε μελέτη οικονομικών επιπτώσεων τη πρόταση αυτή. Θα γίνει στα τέλη του έτου, γιατί είπαμε ότι θα στείλουμε τα αποτελέσματα αυτού του πειράματο στην Επιτροπή και τα κράτη-μέλη κατά τι αρχέ του επόμενου έτου, άρα θα πρέπει να κάνουμε την αξιολόγηση στα τέλη του τρέχοντο έτου. Και έρχομαι στο δεύτερο παράδειγμα, στο δεύτερο διάταγμα που σας ανέφερα, που είναι ένα σχέδιο διατάγματος για την αναφορά χώρα προέλευσης ε, κρέατος ε, και ε, ψαριού όταν χρησιμοποιούνται σε, ως συστατικά σε γεύματα μαζικής εστίασης. Και έτσι είτε πολλούνται σε καντίνα, σε νοσοκομείο, σε σχολείο, αλλά κυρίως σε εστιατόρια, αν χρησιμοποιούνται κρέας ε, ή ψάρια στα γεύματα αυτά και, και αλλά δεν μιλούμε για όλα τα προϊόντα, μάλλον για ορισμένα προϊόντα. Αν όμως έχουμε μία μερίδα που έχει ψάρι ή κρέας, θα πρέπει να αναφέρεται η κρεας θα πρεπει να αναφέρει την προελευση του ψαριού του κρέατος. Και θα πρέπει η μνή αυτή να γίνεται γραπτός, ώστε να μην βάλουμε σε πειρασμό τον ε, παραγωγό του προϊόντος του προμαθευτή του προϊόντος να παραπληροφορεί τον καταναλωτή ή να δίνει ανακριβείς πληροφορίες. Δυστυχώς ήταν αρνητική η αντίδραση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για το διάταγμα αυτό, όπως φάνηκε το Φεβρουάριο φέτος, με την αρνητική γνωμοδότηση, ε, με διάφορους λόγους που επικαλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αρνητική της γνώμη. Πάντως, ε, σημειώνουμε και λαμβάνουμε υπόψη τα προβλήματα που μας επισήμενε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είτε τον Ιούνιο είτε τον Ιούλιο θα υποβάλλουμε νέο διάταγμα. Ε, ε, μάλιστα σκεφτήκαμε να είναι διαιτής η διάρκεια και του δεύτερου διατάγματος γιατί ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι κατά της απεριόριστης εφαρμογής, θέλει χρονικό οριοθετημένο διάταγμα και είχαμε δηλώσει ότι το διάταγμα αυτό θα φορά κάθε είδους κρέας και ψάρι, αλλά ε, θα το περιορίσουμε τελικά σε ορισμένα προϊόντα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ε, ρώτησε αν όντως οι καταναλωτές θεωρούν ως στοιχειοποιότητας ε, την ε, περιοχή, τη χώρα προέλευσης. Εμείς, ε, μάλλον αφελώς, παρουσιάσαμε το ενδιαφέρον των ε, καταναλωτών να περιστρέφεται γύρω περισσότερο από την καλή μεταχείριση των ζώων, την ευζοία ή την ασφάλεια των τροφίμων. Αλλά θεωρούμε ότι πολλοί Φιλανδοί καταναλωτές θεωρούν ότι τα φιλανδικά τρόφιμα είναι ασφαλέστερα. Αυτό όμως δεν το δέχτηκε και πολυθετικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι επαρκής και όλα τα ευρωπαϊκά τρόφιμα είναι εξορισμού ασφαλή. Οπότε θα το λάβουμε αυτό υπόψη για το μέλλον και στη συνέχεια θα χρησιμοποιούμε μόνο το επιχείρημα της ποιότητας. Πάντως θεωρούμε ότι και το σχέδιο διατάγματος είναι καλό γιατί στα εστιατόρια κυρίως οι καταναλωτές ε, παραπλανούνται, ε, ξεγελιούνται και μερικές φορές ε, καταναλώνουν φαγητό ημερίδες που δεν προέρχονται από εκεί που νομίζουν οι καταναλωτές ότι προέρχονται. Γιατί πολλές φορές εισαγόμενο κρέας ψάρι περιλαμβάνονται σε προϊόντα μαζικής εστίασης, όχι τόσο σε αυτά που αγοράζουν τα νοικοκυριά. Δεν είναι προστα απογοητευτικό αυτό το διάταγμα. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που ίσως ε, να φαίνεται να προωθούν ε, την εσωτερική αγορά, αλλά για μας που είμαστε μια σκανδιναβική χώρα, ε, η διαφάνεια είναι σημαντικό ζητούμενο και πρωταρχική μας προτεραιότητα. Θέλουμε να δίνουμε όλες τις, όλες τις πληροφορίες στον καταναλωτή για τον ενημερώνουμε πλήρως. Και σίγουρα η χώρα προέλευσης είναι ένα θέμα που θα πρέπει να γίνεται γνωστό. Θα πρέπει ο καταναλωτή να γνωρίζει από πού προέρχεται ε, το βασικό συστατικό ή το συγκεκριμένο τρόφιμο. Και το ζητούμε αυτό ως ε, νομοθέτες. Γιατί λοιπόν να μην δίνουμε αυτή την πληροφορία και στου καταναλωτές που ή άλλως τη θέλουν. Επίσης, ε, δεν είναι όλα φυσικά τόσο κατηγορηματικά, τόσο άσπρο-μαύρο. Νομίζω ότι σε όλες τις χώρες οι καταναλωτές δεν αγοράζουν μόνο εγχώρια προϊόντα. Μερικές φορές ε, εσκεμμένα αγοράζουν εισαγόμενα προϊόντα, ίσως επειδή είναι πιο ευαισθητομένοι σε θέματα ε, καλής μεταχείρισης είτε για άλλο θέμα. Δεν είναι μονόδρομος λοιπόν, είναι αμφίδρομη διαδικασία, αλλά θα, γι' αυτό ακριβώ θα πρέπει ο ε, καταναλωτής να γνωρίζει και να μπορεί περιστατωμένα να κάνει την επιλογή του και κατατοπισμένα πριν την κατάρτιση του διατάγματος φυσικά εξετάσαμε την άποψη και των καταναλωτών και το 2015 εκπονήσαμε μια ευρύς κλίμακος ε, μελέτη στην οποία διαπιστώσαμε ότι 90% των καταναλωτών στη Φιλανδία ενδιαφέρονται για την προέλευση των προϊόντων των τροφίμων τους. Και στην τελευταία ε, δημοσκόπηση πάλι είχαμε σημαντικό ποσοστό. Και στην πρόσφατη μελέτη του Μαΐου, 82% των καταναλωτών δήλωσαν ικανοποιημένοι από το περσινό διάταγμα. Και εδώ εξετάζουμε το διάταγμα που δεν πέρασε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το τελευταίο ποσοστό είναι το 82% που είναι ο αριθμός των καταναλωτών που πιστεύει ότι θα πρέπει να έχουν γραπτές πληροφορίες για την πρέλευση των τρόφιμων στα ε, τρόφιμα που καταναλώνουν στα εστιατόρια, στους χώρους μαζικής εστίασης. Αυτά ευχαριστώ και θα παραμείνω και στη συνέχεια για τη συζήτηση. Πολύ ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Χέλμ. Περνάμε στην τρίτη παρουσίαση ε, που είναι η παρουσίαση της κυρίας Πέχα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Καταναλωτών. Δέκα λεπτά και εσείς παρακαλώ. Θα τα πω στα γαλλικά διότι θα μιλήσω για το γαλλικό πείραμα μετά από έρευνα που έγινε. για τη ε, γαλλική ε, νομοθεσία. Πρώτα όμως για την οργάνωση που εκπροσωπώ, την ΜΠΕΚ, το Ευρωπαϊκό ε, Γραφείο Πρόσθεσης του Καταναλωτού. Είμαστε Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία, εκπροσωπούμε 43, 43 οργανώσεις, με στόχο να μεταφέρουμε τις απόψεις και να εκπροσωπούμε τα συμφέροντα των καταναλωτών ε, στις, ε, ε, στα ευρωπαϊκά επίπεδα και θεωρούμε ότι οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν την προέλευση των τροφίμων που καταναλώνουν. Το ερώτημα αρχικά δεν είναι και τίποτα το νέο για το και γιατί δουλεύουμε για πολλά χρόνια επάνω σε αυτό. Το από το 2012 είχαμε αναθέσει μια μελέτη σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες Αυστρία, Γαλλία, Σουηδία και Πολωνία μελέτη για να αξιολογηθούν οι προσδοκίες των καταναλωτών σχετικά με την προέλευση. 70% κατά μέσον όρο των καταναλωτών επιθυμούν να γνωρίζουν την προέλευση των τροφίμων. Είναι σημαντικό κριτήριο επιλογής για αυτούς. Πιο πολύ για το κρέας, 90% των καταναλωτών θέλουν να γνωρίζουν την προέλευση του κρέατος που ε, καταναλώνουν, άλλα προϊόντα όπως τα ψάρια, τα φρέσκα λαχανικά, μετά το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου πάλι εκεί άνω των 90% ή άνω των 80% των καταναλωτών επιθυμούν να γνωρίζουν την προέλευση των προτροφίμων αυτών. Άλλο, άλλη πληροφορία που προέκυψε από τη μελέτη είναι ότι θέλουν να γνωρίζουν την χώρα, αν όχι και την περιφέρεια από την οποία προέρχεται Δηλαδή ε, απλώς τα δύο ε, Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τους αρκεί, τουλάχιστον για αυτούς που ερωτήσαμε. Τέλος, το τελευταίο βασικό ε, θέμα είναι ότι ετικέτες για την ώρα, οι επισημάνσεις δηλαδή, δεν τους αρκούν. Θέλουν να γνωρίζουν και που γίνεται η μεταποίηση του προϊόντος, αλλά κυρίως η προέλευση των πρώτων υλών. Μετά από τη μελέτη αυτή, διεξαγάγαμε εκστρατεία μεταξύ 2014-2016 σχετικά με το κρέας, τον οπό κρέας αλλά και το μεταποιημένο. Και βρήκαμε απήχηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύο φορές ψήφισε ψηφίσματα με μεγάλη πλειοψηφία για την υποχρεωτική επισήμανση του νοπού κρέατος αλλά και του μεταποιημένου κρέατος όποτε χρησιμοποιείται δηλαδή σε άλλα τρόφιμα. Δεν ακολουθήθηκαν τα ψηφίσματα αυτά από ευρωπαϊκές δράσεις Γι' αυτό παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα εθνικά μέτρα που λήφθηκαν σε ορισμένε χώρε μέλη, όπω στη Γαλλία. Λίγα λόγια για την γαλλική αντίδραση με διάταγμα του 2016 το οποίο διάταγμα υποχρώνει τους ε, παραγωγούς και τους βιομηχάνους να αναφέρουν την προέλευση του κρέατος εφόσον είναι άνω του 8% του προϊόντος όπως προϊόντα κρέατος, ε, έτοιμα φαγητά κλπ. Υποχρεώνει επίσης τους ε, επαγγελματίες ε, να αναφέρουν την προέλευση του γάλακτος όταν αυτό αποτελεί μέρος το τροφίμου πάνω του 50% και κυρίως δηλαδή για όρθια, τυριά, κρέμες κλπ. Σε ό,τι αφορά το κρέας πρέπει να αναφέρεται η χώρα γέννησης του ζώου, εκτροφής του και σφαγής του. Και Αλλιώς μπορούν να αναφέρονται πιο γενικές πληροφορίες όπως Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Το ίδιο για το γάλα που χρησιμοποιείται ως συστατικό του τροφίμου. Αρκεί να αναφέρεται το σημείο συλλογής του γάλακτος και μετά τη μεταποίηση του τελικού προϊόντος. Και εκεί υπάρχει κάποια ευκαμψία στην περίπτωση όπου αυτές, τα διαφορετικά αυτά στάδια ε, λαμβάνουν χώρα σε διαφορετικές χώρες μέλη. Πρόκειται για ένα διάταγμα το οποίο θα ισχύσει μέχρι τέλους του έτους και μετά θα υποβληθεί έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις ε, επιπτώσεις. Και πρόκειται και για στοιχείο αμοιβαίας αναγνώρισης Δηλαδή το μέτρο εφαρμόζεται μόνο στους παραγωγούς οι οποίοι παράγουν σε γαλλική επικράτεια. Αυτό που μας ενδιαφέρει να μάθουμε είναι αν είχε θετικό αντίκτυπο το μέτρο αυτό στους καταναλωτές. Προσπαθήσαμε να αξιολογήσουμε μέσω ερευνών, πρώτον το 2016 και μετά το 2018. Πριν όμως να γίνει η μελέτη αυτή, είχαμε 244 μεταποιημένα προϊόντα και είχαμε διαπιστώσει τότε ότι δεν μπορεί κανείς να επαφίεται στην βούληση των ε, βιομηχάνων για να δώσουν περισσότερη διαφάνεια στους καταναλωτές σε ό,τι αφορά την προέλευση του προϊόντος και ιδίως του κρέατος. Δεύτερη έρευνα στις αρχές του τρέχοντος έτους για 269 προϊόντα, 53 γαλακτομικά και 216 που περιέχουν και κρέας και για να μπορέσει να γίνει η σύγκριση και η ενδεχόμενη, να μελετηθεί η ενδεχόμενη εξέλιξη αναφέρθηκαν σε όσα είχαν κάνει αναλύσει ήδη το 2016 και αυτό που διαπιστώθηκε είναι ότι αυτοί που ενδιαφέρονται για την προέλευση μετά από τη νέα γαλλική νομοθεσία το αποτέλεσμα ήταν πολύ θετικό για τον γαλακτοκομικό τομέα διότι 89% των προϊόντων που, έχουν, που ανέλησαν αναφέρουν την επισήμανση αναχώρα η χρήση ε, χαρακτηριστικών προελεύσεως γενικότερων όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. κυρίως για κρέας κοτόπουλου και χοιρινού. Ένα μεγάλο ποσοστό δεν περιλαμβάνει τίποτα, αλλά δεν είναι προφανές αν πρόκειται για παραβίαση ή αν πρόκειται για προϊόν το οποίο έχει ε, παραχθεί εκτός της γαλλικής επικρατείας. Τώρα, για πιο λεπτομερή ανάλυση, την αναφορά της προέλευσης ανακατηγορία προϊόντων, γαλακτοκομικών και κρέατος έχουμε επιβεβαίωση των προηγούμενων ε, αξιολογήσεων, δηλαδή με εξαίρεση το γάλα, το γάλα και το ε, τυρί, το 80% αναφέρεται. Για το κρέας είναι πιο διαφορετικά τα πράγματα, διότι αναφέρονται κυρίως εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης παραγωγή, ιδίως για σαλάτες κλπ. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της ε, δήλωσης προέλευσης 2016-2018 κυρίως πάλι για τα προϊόντα κρέατος, διαπιστώνουμε και πάλι ότι η επίπτωση του γαλλικού μέτρου ήταν πολύ θετική και κρίθηκε πολύ ευνοϊκά από τους καταναλωτές για την προέλευση του κρέατος. Ενδιαφέρονται για προϊόντα που το 2016 δεν ανέφεραν καμία, δεν καμία αναφορά προέλευσης ενώ τώρα 60% έχουν. Το ίδιο για τα προϊόντα που το 2016 ανέφεραν μόνο Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, 27% έχουν τώρα πιο συγκεκριμένες αναφορές προέλευσης. Ποιες πληροφορίες μπορεί να αντλήσει κανείς από τις μελέτες αυτές. Πρώτα, ότι τα γαλλικά μέτρα έχουν σημαντική θετική επίπτωση στους καταναλωτές για τα γαλακτοκομικά πάντα και για το κρέας. Αύξηση δηλαδή της ε, διαφάνειας κατά 25% διότι προϊόντα που το 2016 δεν είχαν καθόλου ε, επισήμανση ή πολύ γενικές επισήμανσεις. Τώρα αυτά, ε, το ποσοστά αυτά έχουν αυξηθεί σημαντικά. Έγινε προσπάθεια Σύγκριση των πρακτικών με χρήση τεχνικών στοιχείων για την αύξηση της διαφάνειας. Πρόκειται όμως πραγματικά για πολιτική των επιχειρήσεων. Πιο θετική απέναντι στην διαφάνεια. Θα πρέπει εκεί να τύχουν και οι παραγωγοί καλή θέληση. θα πρέπει να είναι πιο ορατά όταν πρόκειται για σκοπούς marketing. Αυτό που διεπίστωσαν επίσης είναι ότι για προϊόντα που στο πακέτο επάνω να φέρουν με μικρά γράμματα εκτός ή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκεί είναι πολύ πιο... Έχει διαφοροποιηθεί αυτό, γράφουν για παράδειγμα ότι έχει παραχθεί στην Γαλλία. Ότι ένα στάδιο πάντως της παραγωγής έχει γίνει στην Γαλλική επικράτεια. Τώρα, οι συστάσεις του, της οργάνωσης μας BERC θεωρούμε ότι εξακολουθεί να υπάρχει πολύ έντονη επιθυμία από τους Ευρωπαίους καταναλωτές να γνωρίζουν την προέλευση ιδίω του κρέατος και των γαλακτοκομικών προϊόντων είτε ε, αστούσιων είτε ω συστατικών τροφίμων. Υπάρχει το άρθρο 26 παράγραφος 3 που αναφέρθηκε προηγουμένως αλλά δεν θεωρείται ότι αρκεί διότι αναφέρεται μόνο στις περιπτώσεις όπου οι παραγωγοί αποφασίζουν εθελοντικά να παράσχουν τις σχετικές ε, πληροφορίες. Και τέλος, συνεχίζει τη συζήτηση και ελπίζουμε ότι οι διάφορες εκθέσεις που θα προέρχονται από τις χώρες μέλη που έχουν κάνει ε, τις πειραματικές, τα πειραματικά αυτά μέτρα θα βοηθήσουν ώστε να προαχθεί. Είμαι στη διάθεση σας για ερωτήσεις. Ευχαριστούμε θερμά τους εμπειρογνώμονές μας για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις που μας έκαναν και ο συνήθως θα ακολουθήσει συζήτηση προκειμένου να ευλουτίσουμε ακόμη περισσότερο τις γνώσεις μας. Ο κύριος Αντεκάστρο πρώτος. Δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλου του φιλοξενούμενου μα τη απογευματινή συνεδριάσεω. Η παρουσία ήταν άκρο ενδιαφέρουσα. Να υπενθυμίσω μόνο πώ μετά τα διάφορα πειράματα που έγιναν στην Ευρώπη, αν θυμάμαι σωστά, οκτώ χώρε εφάρμοσαν εθνικές προδιαγραφές για την ετικετοθεσία προέλευσης Προφανώς, συνάδελφοι, επιβάλλεται μια αναθεώρηση της βασικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Να υπενθυμίσω σε όλους τους συναδέλφους σήμερα. Ο Μάρκ Ταραμπέλα έφυγε. Ο Μάρκ Ταραμπέλα είχε ετοιμάσει γνωμοδότηση Επιτροπής Γεωργίας στην προηγούμενη θητεία και προτείναμε τότε την έκθεση Σόμερ που έγινε ο κανονισμός ο βασικός όσον αφορά την ετικεταθεσία. Είχαμε προτείνει υποχρεωτική αναφορά προέλευσης για όλα τα τρόφιμα αναφέροντας τον καταναλωτή σαφώς την προέλευση του βασικού στατικού του τροφίμου. Ερώτηση. Αυτή η εφαρμοστική πράξη που ο Επίτροπος Ανδρουκάητης παρουσίασε πριν από κάποιες εβδομάδες που αναγνωρίζει βέβαια, αναγνωρίζουμε ότι κάνει σημαντικά βήματα πρόοδου όσον αφορά τον υποχρεωτικό χαρακτήρα μόνο στην περίπτωση όπου υπάρχει ένδειξη στην ετικέτα να υπάρχει αναφορά της χώρας η, η υπενθύμηση συγκεκριμένης χώρας όμως προφανώς αυτό το μέτρο δεν επιτρέπει το να επανεξετάσουμε το βασικό κανονισμό ούτω ώστε στην επόμενη θητεία να υπάρχει δυνατότητα να θεσπιστεί μια νομοθεσία που ζητούν και οι κατανοτές ευρωπαϊκών χωρών αλλά και εμείς στην Ολομέλεια, στο Ευρωκοινοβούλιο. Επανειλημμένα ζητήσαμε. Το υπενθύμησε ένα φιλοξενούμενο. Πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορούμε να ενστερνιστούμε αυτό το στόχο και να το προτείνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Γιλέρα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους καλεσμένους μας για τις ομιλίες τους. Μας παρουσίασαν τις ε, εθνικές πρωτοβουλίες στις χώρες τους. Κάτι που μου τράβηξε την προσοχή είναι το εξή. Ε, ναι, μεν έχει νόημα η επισήμαση της χώρας προέλευσης, κυρίως για να κατατοπίζονται οι καταναλωτές, αλλά αν αυτό επιπλέον όπως είπε ο κύριος Μονκάλβο, έχει θετική απήχηση και στους παραγωγούς, τόσο το καλύτερο. Γιατί είπατε ότι αυξήθηκε κατά 25% η αξία σε επίπεδο παραγωγού, ε, κτηνοτρόφου ή γαλακτοπαραγωγού και μάλιστα οδήγησε και στην αύξηση της τιμής του προϊόντος. Οπότε ενώ βελτιώθηκε η τιμή παραγωγού, ε, η τιμή δηλαδή για τους ε, γαλακτοπαραγωγούς, ε, δεν αυξήθηκε η τελική τιμή του προϊόντος, οπότε είναι προ όφελο και των παραγών και των καταναλωτών. Και αν όντω έχουμε τέτοια αποτελέσματα με την επισήμανση, τόσο το καλύτερο. Αυτό ήταν το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που συγκράτησα από τι παρεμβάσει. Αυτό που με προβληματίζει είναι το εξή. Εγώ είμαι υπέρ τη επισήμανση. Η κυρία Περά μα παρουσίασε την γαλλική περίπτωση. Εγώ φοβάμαι μήπως ε, έχει κάποια, ε, κάποιο απόϊχο προστατευτισμού αυτή η διάταξη. Ναι, είναι ενδιαφέρον αυτό, αυτή η απέτηση των καταναλωτών και το μέλημα της διαφάνειας. Αλλά η προέλευση ε, δεν δίνει στοιχεία ούτε για το μοντέλο παραγωγής, ούτε για την τήρηση των διατάξεων της ε, καλής μεταχείρισης των ζώων. Απλώς αναφέρεται στην εγκύτητα. Οπότε το... είναι ενδιαφέρον αυτό το διτό παράδειγμα και ίσως θα μπορούσαμε στην επόμενη κοινοβουλευτική θητεία να εξετάσουμε ακόμη και μεταρρύθμιση νομοθεσίας, αλλά αυτό που με προβληματίζει είναι να μην εκτραπούμε προς κάποιον προστατευτισμό και πώς μπορούμε να αποφύγουμε κάτι τέτοιο, να ε, μπέσουμε σε προστατευτισμό. Να περιπέσουμε σε προστατευτισμό. Κύριε Σαντρία, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συνεχίζω το λογικό ήρμο των προελισσάντων και θα ήθελα φυσικά να σας ευχαριστήσω και να πω ότι από τις τρεις παρουσιάσεις προέκυψε η ανάγκη αναθεώρησης της σχετικής νομοθεσίας το οποίο έχουμε ζητήσει επαγγελμένο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχω λοιπόν μία ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ερωτήσεις προς τους εμπειρογνώμονες έχουμε κάποια αξιολόγηση που γίνεται όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δούμε τι συνέπειε αυτών των τριών εθνικών πειραμάτων. Θα ήταν πολύ σημαντικό να γίνει μια τέτοια αξιολόγηση και θα προκαθορίσει και τι μελλοντικέ μα ενέργειες. Αυτό προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, ως προς τις εθνικές διατάξεις. Ε, ε, η προέλευση, η επισήμανση προέλευση είναι ε, απαραίτητος όρος, αλλά όχι ικανός, ικανή προϋπόθεση, επαρκής προϋπόθεση ε, για να ικανοποιήσουμε τις απαιτήσει των καταναλωτών για διαφάνεια. Θα πρέπει στο μέλλον να λάβουμε υπόψη και άλλα στοιχεία πέραν της προέλευσης. Επίσης, είχαμε αύξηση του κόστους για τους ε, προμηθευτές τροφίμων στην τροφική αλυσίδα. η επισήμανση είχε σημαντικές συνέπειες στον ανεφοδιασμό και Χρειάστηκε παραγωγή παραγωγή να προσαρμόσουν τα στήματα παραγωγής του, ώστε να κάνουν μία διάκριση των προϊόντων ανάλογα με την προέλευσή τους. Οπότε κάτι τέτοιο είχε κάποια επιβάρηση κόστους για αυτούς. Επίσης, η ετικετοθεσία αυτή οδήγησε σε κατακαιρματισμό των εμπορικών συναλλαγών στην, Ευρω... στην ενιαία αγορά. Αυτά είναι τα τρία στοιχεία, τρεις απορίες μου και θα ήθελα περισσότερες λεπτομέρειες με βάση τα τρία εθνικά πειράματα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντόρφμαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πάνω σε αυτά που είπε ο Παύλο Κάστρο. πρώτα απ' όλα θα πρέπει να εξετάσουμε του ευρωπαϊκούς κανόνες αν χρειάζεται να είναι πιο ακριβή όσον αφορά την αναφορά προέλευσης των προϊόντων. Είναι και θέμα εσωτερική αγοράς στην Ευρώπη. Έχω δύο ερωτήσει που θέλω να απευθύνω στο πάνελ. Είναι σαφές ότι οι καταναλωτές στον τομέα της διατροφής, όταν ζητάμε τι θέλει, δεν θέλει ο καταναλωτής, πολύ συχνά δεν λέει την αλήθεια ο καταναλωτής. Καμιά φορά λέει λίγα. Υπάρχουν μελέτες, ρωτήθηκαν οι καταναλωτές αν πραγματικά έλεγξαν την ακρίβεια αυτών που αναφέρονται στη συμβασία του γάλακτος ρωτήσανε στην υπεραγορά. Εσύ, εσύ όταν αγόρασες από το ράφι τη συσκευασία του γάλακτος ή το γιαούρτι, το εξέτασες, εξέτασες την ε, ετικέτα. Ίσως θα ήταν διαφορετικά τα στοιχεία για τους ελέγχους. Αυτό το σύστημα λειτουργεί ανελέγχεται. Για τις χώρες αυτές ποιο είναι το ελεκτικό σύστημα σήμερα. Υπάρχει ένα σύστημα ελέγχου που εφαρμόζεται και πώς λειτουργεί το σύστημα ελέγχων. Ευχαριστώ κύριο ähm, äh, äh, Ευχαριστώ για τι παρεμβάσει σα. Έχω διάφορε ερωτήσει, γιατί αυτά ενδιαφέρουν και του ε, γαστρονόμους εστιατόρε δηλαδή κλπ. βεβαίω και του καταναλωτέ. Είπατε ότι στην Ιταλία αυξήθηκαν οι τιμές κατά 25%. Όχι όμως η τιμή του καταναλωτού. Είχε πέσει τότε όμως η τιμή του καταναλωτού. Όταν είχαν πέσει οι τιμές. Από όσο ξέρω μόνο 6% του γάλακτος φτάνει στα ράφια ως νοπό γάλα. Αυτό ίσως έχει ενδιαφέρον. Και τελευταία ερώτηση. Όταν ένας χείρος έχει εκτραφεί με 90% ε, σόγια ή ε, άλλες ζωοτροφές από τις ΗΠΑ ή τη Βραζιλία. Θεωρείται ακόμα ότι πρόκειται για γαλλικό ή ε, φιλανδικό χείρο κλπ. Κύριο Σάγνιου, είναι επανάσταση θα έλεγα όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για περισσότερη ετικετοθεσία που θα αναφέρεται η χώρα παραγωγής του τροφίμου. Σε έναν ευρωπαϊκό ιδεώδη κόσμο, όλα αυτά είναι ευρωπαϊκά τρόφιμα. Δεν θα έπρεπε να μα προβληματίζει αυτό. Διότι θα εξαφανιστούν τα κράτη-μέλη με την πάω του χρόνου. Ποιο είναι το πρόβλημα όμω. Οι αιρετοί εκπρόσωποι της, του λαού έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι αιρετοί εκπρόσωποι βρίσκονται εδώ και οι γεωργοί μας λένε ότι πρέπει να τους βοηθήσουν. διότι έχουμε κακές τιμές. Κοιτάξτε όλο το εισαγόμενο τρόφιμο που έρχεται από γειτονική χώρα. Αν δεν ερχόταν αυτό, θα είχαμε υψηλότερε τιμέ, λένε οι Γεωργοί. Οι γειτονικέ χώρε πιθανότατα είναι χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε οι αιρετοί εκπρόσωποι έρχονται εδώ για να αντιταχθούν στην έννοια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω να καταλαβαίνετε το πνεύμα μου. Πάντα είχαμε αυτή την ανησυχία στον Ηνωμένο Βασίλειο θα θέλαμε να τονίσουμε κάτι και να πούμε αυτό είναι καλό διότι είναι βρετανικό, αλλά δεν μα επιτρέπεται να το κάνουμε αυτό και το κανόνα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Οπότε έπρεπε να φεύγουμε ένα σύστημα, το, ρε, το κόκκινο τραχτέρ, όπου ενθαρρύνουμε του παραγωγού να συμμορφωθούμε κάποιε προδιαγραφέ και ενθαρρύνουμε τι υπεραγορέ να αγοράσουν αυτού που παράγουν τα προϊόντα και εφόσον είναι μόνο Βρετανοί παραγωγοί που συμμορφώνονται και παράγουν σε αυτά τα πρότυπα, προσπαθούμε αυτό να παραμείνει εντό του οίκου. Έτσι το υπερκεράσαμε το πρόβλημα. Υπάρχουν τριών ειδών καταναλωτές. Εκείνοι που αγοράζουν βάσει τιμής. Αυτό τους ενδιαφέρει, μόνο η τιμή. Υπάρχουν εκείνοι που θα υποστήριζαν τη χώρα τους εάν μπορούσαν και θα συγχωρούσαν κάποια χρήματα παραπάνω εάν μπορούσαν να στηρίξουν τους γεωργούς αλλά δεν μπορούν να το διαπιστώσουν. Και μετά έχουμε τους άλλους που αγοράζουν για άλλους λόγους. Ότι είναι βιολογικό προϊόν ή είναι στα πλαίσια του δικαίου εμπορίου. Τι θα συμβεί εδώ. Θα δούμε μια μετακίνηση από τιμή προς χώρα επιλογή βάση τη χώρα. Κυρία Γκοσέφσκα, ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους καλεσμένους μας ε, για τις παρουσιάσεις της. Ε, μια και έχουμε λίγο χρόνο, θα ήθελα να αναφέρω κάτι που ε, αναφέρεται πολύ συχνά στον πολωνικό τύπο, ότι οι και πατάτες, γερμανικά γιαωμήλα, πολλούνται στην Πολωνία ως πολωνικά τρόφιμα. Και μάλιστα η παραγωγή λένε από τη στιγμή που η απολύμαση έγινε με πολωνικές προδιαγραφές στην Πολωνία μπορούν να χαρακτηρίζονται ως πολωνικά προϊόντα. Ε, ενώ κανονικά θα έπρεπε να αναφέρεται στην επισήμαση χώρα προέλευσης Γερμανία και όχι η Πολωνία. Μερικές ε, εταιρείε κάνουν κατάχρηση της κατάστασης και μπορούν να χειραγωγήσουν με παραπληροφόρηση τον καταναλωτή. Ευχαριστώ. Δεν ζητάει άλλος κανείς το λόγο. Οπότε θα δώσω το λόγο στους καλεσμένους μας για να απαντήσουν σύντομα στις απορίες των Ευρωβουλευτών. Δύο λεπτά ο καθένας επίσης όπως και τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας. Μα τη σειρά που μιλήσατε και προηγουμένως αν θέλετε. Okay. Θα προσπαθήσω να διατρέξω όλες τις ερωτήσεις. Όσον αφορά την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των διαταγμάτων. Όσον αφορά την Ιταλία, το διάταγμα για την προέλευση του γάλακτος σε όλα τα προϊόντα τα παράγωγα του γάλακτος που ετέθησε ισχύ Απρίλιο 2017 με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βλέπει επαλήθευση μετά από δύο χρόνια τη πειραματικής εφαρμογή, όπω προβλέπεται και από τον κανονισμό το 1169. Σε αυτή τη φάση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ακόμα εμβαθύνει στα αποτελέσματα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του Ιταλικού διατάγματος, ενώ το Ιταλικό Υπουργείο και οι φορείς οι ελεγκτικοί της αγοράς στην Ιταλία κάνουν τις αξιολογήσεις τους. Το στοιχείο όσον αφορά την αύξηση των τιμών του γάλακτος και στην εκμετάλλευση και στην κατανάλωση που σας έδωσα αυτά τα στοιχεία είναι στοιχεία που προέρχονται από τις αναλύσεις του Υπουργείου. Το φορέ του Υπουργείου που ασχολείται με τον έλεγχο των τιμών, το ΙΣΜΕΑ, μαζί με την Ένωση Nielsen, την εταιρεία Nielsen, έκαναν δημοσκόπηση τη αγορά το πρώτο έτος εφαρμογής και έτσι είδαμε κάποιες ενδείξεις όσον αφορά την τιμή του γάλακτος στην κατανάλωση που όπως έλεγα αυξήθηκε μόνο κατά 0,6% και ανάλυση όσον αφορά τις τιμές των ε, φτηριών δεν δείχνει αυξήσεις ε, υπέρμετρες στα άλλα προϊόντα γάλακτος. Αυτή η αύξηση του 25% της τιμής στην εκμετάλλευση, στην παραγωγή στην περίοδο μεγάλης κρίσης που αντιμετωπίζει το Ιταλικό γάλα και το γάλα σε πολλές χώρες Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκή έγινε και λόγω της, ήταν αποτέλεσμα και τη κυριοθεσία. Και αυτή η βελτίωση της τιμής καταφέρνει να παραμένει και σήμερα. Όταν δυστυχώς υπάρχουν σήμερα διάφορα μηνύματα υποχώρησης της οικονομίας σε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όσον αφορά την προέλευση, αν είναι αναγκαίο ή αρκετό. Η προέλευση είναι σημαντικό βήμα, διότι είναι ουδέτερη πληροφορία που επιτρέπει επιλογή στους πολίτες. Δεν θέλουμε να σπρώξουμε τους πολίτες να επιλέξουν το προϊόν της χώρας τους, του κράτους μέλους τους. Θέλουμε να δώσουμε ουδέτερες πληροφορίες που επιτρέπουν στους πολίτες να επιλέξουν. Σίγουρα θα υπάρξουν πολίτες που θα αγοράσουν κυρίως προϊόντα της χώρας τους, αλλά οι έρευνες της αγοράς μας επιβεβαιώνουν ότι δεν κάνουν όλη αυτή την επιλογή με βάση εθνικιστική. Αλλά είναι ουδέτερη ενημέρωση στην ετικέτα που χορηγείται και είναι πληροφορίες αυτές που δίδονται σημαντικές. Οι καταναλωτές προφανώς ζητούν περισσότερα από μας, θέλουν να ξέρουν περισσότερα ποια είναι τα επίπεδα βιωσιμότητας, περιβαλλοντικής, ευημερίας των ζώων και σεβασμού των εργαζομένων που χρησιμοποιούνται στις εταιρείες παραγωγής της γεωργικές. Και αναφορά προέλευσης της χώρας επιτρέπει στους πολίτες να ε, εξετάσουν ποιοι είναι οι κανόνες που ισχύουν εκεί, ποια είναι η νομοθεσία με την οποία συμμορφώνονται οι γεωργοί εκεί. όμως αυτό που ανησυχεί περισσότερο είναι τα συστήματα ετικετοθεσίας επιθελοντικής βάσης για την ώρα, όπως η ετικέτα με κάποιο σήμα που εφαρμόζεται, με κάποιο σήμα χρώμα, όπως σε κάποιες ευρωπαϊκές, ε, αγγλικές ευρω... Ε, υπεραγωγές ή στο, ε, στα γαλλικά σούπερ μάρκετ. Δεν είναι ουδέτες πληροφορίες, αλλά μέσα αυτού του σήματος προσπαθούν να παρασύρουν τον καταναλωτή να επιλέξει ένα προϊόν περισσότερο από κάποιο άλλο. Όχι δυνάμει ουδέτερης πληροφόρησης, αλλά μέσω μιας ε, σύνοψης που κάποιος κάνει ή διατείνεται ότι κάνει για να ενημερώσει τον καταναλωτή. Τώρα για τους ελέγχους. Το σύστημα των ελέγχων είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στην Ιταλία όλες οι δυνάμεις της τάξεως που ασχολούνται με τον έλεγχο των τροφίμων ασχολούνται και με την ετικεταθεσία σαν την προέλευση και το κάνει και το Υπουργείο άλλωστε ε, στα πέση καταπολέμηση των απατών. Αύξηση όμω των κυρώσεων που απορρέουν του ελέγχου είναι κάτι πολύ σημαντικό όσον αφορά μόνο την προέλευση του προϊόντο που αναφέρεται υποχρεωτικά, αλλά όλε οι ενδεχόμενε απάτε που διαπράττονται στον τομέα των τροφίμων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Χέλμς από τη Φιλανδία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολλές ενδιαφέρουσες ερωτήσεις, θα προσπαθήσω να απαντήσω με τη σειρά. Για τον κύριο Κάστρο. Συμφωνώ μαζί σας. Στη Φιλανδία πιστεύουμε ότι χρειάζονται ενιαίοι κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι η επισήμαση της χώρας προέλευσης είναι κάτι που θέλουν οι καταναλωτές και το χρειαζόμαστε. Και αν μπορούμε να το επιτύχουμε για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, θα είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση από αυτήν που έχουμε τώρα, όπου έχουμε διαφορετικούς πειραματισμούς σε διάφορες χώρες. Η κυρία Γκασία επίσης έθεσε ένα ενδιαφέρον θέμα για τα συστήματα παραγωγής και ανεξαρτήτως του αν γνωρίζουμε την χώρα προέλευσης, δεν γνωρίζουμε για το σύστημα παραγωγής. Αυτό είναι αληθές. Αλλά νομίζω ότι η χώρα προελεύσεως είναι κάτι εύκολο σχετικά. Δηλαδή βρίσκεται η πληροφορία σχετικά εύκολα. Είναι σαν όριμο φρούτο που κρέμεται. Πιο εύκολο λοιπόν να δώσουμε αυτές τις πληροφορίες. Για τα συστήματα παραγωγής δεν έχουμε πραγματικά συστήματα σε όλες τις χώρες μέλη που να μας επιτρέπουν να γνωρίζουμε ποιο είναι το σύστημα παραγωγής του συγκεκριμένου ε, τροφίμου θα είναι πολύ μεγάλη γραφειοκρατική επιβάρυνση αν ζητήσουμε να γίνει και με τους κανόνες προστασίας των ζώων και με άλλους κανόνες που νομίζω ότι έχουμε εν τέλει συστήματα που μπορεί να μην είναι υποχρεωτικά αλλά δίνουν σποφορές αυτές. Στη Δανία έχουν ένα πολύ καλό ε, σύστημα προστασίας ε, των ζώων και της ευημερίας των ζώων βλέπουν δηλαδή ε, και στη βάση του συστήματος αυτού από όπου προέρχεται το ζώο. Και τέλος το ερώτημα του κύριου Ντόρφμαν για τα συστήματα ελέγχου. Αν δηλαδή έχουμε πράγματι κάποιον τρόπο ελέγχου, άσκηση ελέγχου της επισήμανσης της χώρας προελεύσεως. Και αυτό είναι σημαντικό. Προέρχομαι από τον έλεγχο των τροφίμων. Αν έχουμε πανευρωπαϊκούς κανόνες, πανευρωπαϊκής ισχύω δηλαδή, θα είναι τότε γνωστή σε όλους τους καταναλωτές και οι καταναλωτές έχουν την ικανότητα να διαπιστώσουν αν κάποιος παραπλανά και παραβιάζει τους κανόνες αυτούς. Αν λείπει για παράδειγμα η επισήμανση της προέλευσης. Το βλέπουμε αυτό στη Φιλανδία να συμβαίνει ήδη. Και ε, ο Γερμανός κύριος έθεσε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Αν δηλαδή ο χείρος είναι πράγματι φιλανδικός εφόσον έχει εκτραφεί με βραζιλιάνικο ε, ε, αλεύρι και είναι φιλανδικός ή γερμανικός ή δεν ξέρω τι. Δηλαδή δεν μπορούμε να αποφύγουμε το γεγονό ότι θα χρησιμοποιηθούν διαφορετικά ε, τρό, τρόφιμα για την εκτροφή του, αλλά και η τελευταία φωτογραφία που έδειξα, η τελευταία ε, στην παρουσίασή μου, η τελευταία φωτογραφία έδειχνε ένα γουρουνάκι με ουρά. Και τα χοιρινά αυτά στην Σουηδία και σε εμά είναι τα τελευταία πανευρωπαϊκά που έχουν ουρίτσα. Ε, δεν ξέρω το αν μπορώ αυτό να χαρακτηρίσω το ένα καλύτερο από το άλλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καταρχήν να απαντήσω στον κύριο Τεκάστρο και από τη δική μας κοπιά της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Καταναλωτών είμαστε υπέρ πανευρωπαϊκών κανόνων για την, ε, για την ε, αναφορά της χώρας προέλευσης γιατί εξασφαλίζουμε ισότιμη πληροφόρηση όλων των καταναλωτών. Αυτό ελπίζω να είναι προτεραιότητα και στο επόμενο κοινοβούλιο κάτι τέτοιο. Σε ό,τι φορά το σχόλιο της κυρίας ε, Αγγιλέρα κατά πόσο η αναφορά της χώρας προέλευσης ε, συνιστά προστατευτισμό. Όχι κατά τη γνώμη του ΜΠΕΚ της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Καταναλωτών. Αντίθετα δίνει ε, πληροφορίες στον καταναλωτή για την προέλευση του προϊόντος του τροφίμου. Και δεν αναφέρθηκα ούτε σε τρόπο ούτε σε μοντέλο παραγωγής. Πάντως μερικοί μπορεί χρησιμοποιούν το, την αναφορά χώρα προέλευση ω ε, διαφημιστικό εργαλείο όταν ε, του εξυπηρετεί, όταν εξυπηρετεί τη στρατηγική του, ε, όταν θέλουν να προβάλλουν ένα χώριο προϊόν, ένα χώριο συστατικό. Εμεί θέλουμε οι υπεύθυνοι των τροφίμων να δίνουν τι ίδιε πληροφορίε σε όλου του καταναλωτέ, άσχετα με την προέλευση για να μπορούν εμπεριστατωμένοι να κάνουν την επιλογή του οι καταναλωτέ και να διαλέγουν είτε το χώριο προϊόν να το επιθυμούν είτε αν θέλουν να αγοράσουν προϊόν εισαγόμενο να το κάνουν. Είτε επειδή είναι ε, γνωστό, είτε φημισμένο, ε, αλλά τουλάχιστον με διαφάνεια να έχει τις πληροφορίες ο καταναλωτής και να είναι παρόμοιες οι πληροφορίες παντού. Κύριε Ντόρφμαν, υπάρχει μερικές φορές διαφορά μεταξύ των δηλώσεων των καταναλωτών στις δημοσκοπήσεις και της συμπεριφοράς του σε σούπερ μάρκετ. Πάντως, ε, έχουμε διαπιστώσει τη συλλήπεια των καταναλωτών ό,τι αφορά την απέτησή του για τη χώρα προέλευση. Και μάλιστα και σε μελέτε και έρευνε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε ε, έρευνε του Ευρωβαρομέτρου καταλήγουμε στο ίδιο αποτέλεσμα. Ιδιαίτερα για την προέλευση του γάλακτο, αν θυμάμαι καλά, 83% των καταναλωτών δήλωσαν ότι θα ήταν διτεθειμένοι να πληρώσουν ακόμη και υψηλότερη τιμή προκειμένου να έχουν την πληροφορία για τη χώρα προέλευση. Υπάρχει τέτοια προθυμία λοιπόν για τους καταναλωτές Τώρα, αν αυτό χρησιμοποιείται ως εργαλείο ε, για να ε, κρυθεί το αίτημα των καταναλωτών, νομίζω ότι είναι επαρκές εργαλείο. Οι καταναλωτές απαιτούν ενημέρωση για την προέλευση των τροφίμων τους. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε το πρώτο πάνελ της δημόσιας ακροασίας μας. Ακούσαμε τις παρουσιάσεις των καλεσμένων μας εμπειρογνωμόνων. Ε, ακολούθησε και συζήτηση με ερωτήσει από τους ευρωβουλευτές και η εμπειρογνώμονες είχα την ευκαιρία να απαντήσουν και στις ερωτήσεις. Ευχαριστώ θερμά και περνάμε στο δεύτερο πάνελ και καλό τη δεύτερη ομάδα των εμπειρογνωμόνων να λάβει θέση στο Προεδρείο και να καλωσορίσω την κυρία Βαλεάν που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και θα προεδρεύσει στο δεύτερο πάνελ. Παρακαλώ τους εμπειρογνώμονες να λάβουν θέση. Κύριε Αβαλάν, κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Uh, Ευχαριστώ κύριε Σικέρσκι που προεδρεύσατε στο πρώτο πάνελ και που συμφωνήσατε να διαξαχθεί μαζί με την Επιτροπή Περιβάλλοντος αυτή η ακρόαση. Έχω τη τιμή να προεδρεύω του δευτέρου πάνελ που ασχολείται με τομεκή προσέγγιση όσον αφορά την ετικετοθεσία χώρας προελεύσεως, όσον αφορά τα τρόφιμα, ε, το θέμα της ετικετοθεσίας των τροφίμων, κυρίως η ένδειξη προέλευσης, είναι σημαντικότατο θέμα για την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Όχι μόνο διότι είναι ένα τμήμα των αρμοδιοτήτων μας, αλλά διότι συνδέεται στενά με την ασφάλεια των τροφίμων. Ε, πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι απέναντι στου Ευρωπαίου πολίτε, στου καταναλωτέ και έναντι τη υγεία του. Αυτή είναι μια σημαντική πτυχή που προασπίζεται η Επιτροπή περιβάλλοντο, παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς το θέμα και θέλει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα τη απάτη στα τρόφιμα, το θέμα της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα τρόφιμα και το θέμα της λειτουργίας της όλης αλυσίδας διατροφής. Τα δύο ψηφίσματα που υθετήθηκαν στην Ολομέλεια της κατόπιν πρωτοβουλίας Επιτροπής Περιβάλλοντος το 2015 και το 2016 για την ετικετοθεσία για προέλευση τροφίμων στον φωτοκρέας και μεταπημένων τροφίμων και κυρίως για κάποια τρόφιμα αλλά δείχνουν ότι ενδιαφέρεται πολύ το Ευρωκοινοβούλιο για το ζήτημα. Ζήτησαν και τα δύο ψηφίσματα θέσπιση περισσότερων νόμων λαμβάνοντας υπόψη ότι η συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών θέλουν περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την προέλευση των τροφίμων του και την ποιότητά του. Το δεύτερο πάνελ θα εστιαστεί κατά πόσο εφαρμοστικό κανονισμό του 2018 που υιοθετήθηκε πριν από λιγότερο από μία εβδομάδα μπορεί να δώσει σαφήνεια επιτέλου, όσον αφορά το θέμα τη υποχρεωτική ή εθελοντική αναφορά χώρα προέλευση στα τρόφιμα για να προσφέρει διαφάνεια που επιθυμούν οι προβληματισμένοι καταναλωτές και ταυτόχρονα να λάβει υπόψη και αντιμετωπίσει τις ειδικέ ανάγκες και ιδιαιτερότητες των φορέων του τροφιμικού τομέα. Στην προσπάθεια να εξετάσουμε το ζήτημα, σας παρουσιάζω τους τρεις εμπειρογνώμονες. Την κυρία Ντορότα Κοσλόφσκα. Καλώς ήρθατε, Διευθύντρια για θέματα νομοθεσία και των τροφίμων στην Πολωνική Ομοσπονδία του τομέα της των τροφίμων, ο κ. Ντέρκ Ιάκοψ. Καλώς ήρθατε, γεια σας. Υποδιευθυντής της Food and Drink Europe και τον κύριο Παύλο Κάρα, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της International Evasion. Καλώς ήρθατε αφήσαμε για το τέλος της απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η κυρία Αλεξάνδρα Νικόλα Κουπούλου επικεφαλής της μονάδας για την ενημέρωση για τρόφιμα της Γενικής Διευθύνσεως ΣΑΝΤΕ θα μας δώσει κάποιες πληροφορίες όσον αφορά την εφαρμοστική πράξη που εθετήθηκε. Προσβλέπω στη συζήτησή μας, θα υπάρξει και χρόνος για ερωταπαντήσεις στο τέλος των παρουσιάσεων των πάνελ. Να δώσω το λόγο στην κυρία Κοσλόφσκα, Έχετε το λόγο για 10 λεπτά το πολύ. Ορίστε. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι εξότιμοι ευρωβουλευτέ, σα ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας παρουσιάσω την άποψή μας για τον εκτελεστικό κανονισμό 2018-775 και να σα παρουσιάσω τη σκοπιά των επιχειρηματιών που εκπροσωπούνται στην Πολωνική Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τροφίμων ε, που εκπροσωπούν διάφορους κλάδους τροφίμων ε, και επεξεργάζονται προϊόντα με πολλά συστατικά με προορισμό την κατανάλωση. Και πρόκειται για προϊόντα που διατίθεται στην αγορά μέσω λιανικού εμπόριου και αλυσίδων λιανικής διανομής και λιανοπολιτών. Ο εκτελεστικός κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέφθηκε ε, για, για, να, για τον κανονισμό 1169-2011 που προβλέπει την ε, αρχή της ε, αναφοράς χώρας προέλευσης του βασικού συστατικού με βάση το άρθρο 26 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού 1169 του 2011. Δηλαδή, ε, έχουμε την περίπτωση σε που το κύριο συστατικό, το βασικό συστατικό έχει προέλευση διαφορετική από την προέλευση του, του τελικού προϊόντος ε, και μιλούμε για προϊόντα που απαρτίζονται τουλάχιστον από δύο συστατικά. Τώρα, για να μπορέσουν οι επιχειρηματίες να συμμορφωθούν με τον κανονισμό θα πρέπει σε μια πρώτη φάση μετά την ανάλυση του προϊόν, των προϊόντων τους να δουν ε, ποιο είναι το βασικό συστατικό και να, να δουν κατά πόσο αναφέρεται η προέλευση του βασικού συστατικού. Και εδώ μιλάμε για δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Όταν η δήλωση της προέλευσης ε, ήδη παρέχεται υποχρεωτικά από την επιχειρηματία, με βάση το άρθρο 26.2α του βασικού κανονισμού ή αν πρόκειται για εθελοντική αναφορά της προέλευσης. Βέβαια, η περίπτωση των προϊόντων με προστατευμένη γεωγραφική ένδειξη ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα είναι εκτός πεδίου εφαρμογή του εκτελεστικού κανονισμού. Και στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση μελέτε που θα, προ... θα πραγματοποιήσει θα επεκτείνει ενδεχομένω το πεδίο εφαρμογή. Προ το παρόν αποκλείονται όμω. Τώρα, α, είναι σημαντικό ε, να γνωρίζουμε τον ορισμό του βασικού ή κύριου συστατικού. Αυτό είναι σημαντικό και για τους ελεκτικού φορείς. Ε, αυτό με βάση τον ορισμό περιλαμβάνει ο κανονισμό 1169 του 2011. Ο, κανονισμό, ο ορισμός απαρτίζεται από δύο τμήματα. Καταρχήν, ε, ίσως με βάση την ερμηνεία ε, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε διαφορετικό συμπέρασμα για ποια στατικά θα μπορούσαμε να προσφέρουμε τέτοιε πληροφορίε, σε περίπτωση που το, η προέλευση του κύριου στατικού είναι διαφορετική από την προέλευση του τελικού προϊόντο. Γι' αυτό σημαντικό ρόλο έχει ο ορισμό ό,τι αφορά τι δυνατότητε ερμηνεία που παρέχει. Τώρα, ο ορισμός θα πρέπει να είναι άσχετος από τον τρόπο παρουσίασης ε, του τελικού προϊόντος. Μπορεί να είναι ε, δήλωση, μια γραφική παρουσίαση, σύμβολα, όροι ή να αναφέρεται σε μια γεωγραφική περιοχή. Αυτό που είναι ενδιαφέρον για τους επιχειρηματίες και παραγωγούς τροφίμων, ιδιαίτερα τροφίμων που απαρτίζονται από πολλά συστατικά, είναι όταν ε, οι γεωγραφικοί όροι ε, που περιλαμβάνονται σε συνηθισμένα γενικά ονόματα για τα οποία ε, που κανονικά δεν ε, περιέχουν δεν αναφέρουν προέλευση, αλλά κατά την κοινή αντίληψη δεν συλληστούν αναφορά χώρα καταγωγή ή τόπο προέλευση. Στην αγορά υπάρχουν πολλά προϊόντα που στον τίτλο τη αναφέρονται κάποιε προελεύσει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά, την τεχνολογική διαδικασία, την προέλευση, αλλά δεν μιλούν κατά για την προέλευση του, τελικού προϊόντος. Στην πολωνική αγορά ε, είναι πολύ δημοφιλής η, η γκούλας, ε, ουγγρική σούπα. αυτό όμως ε, δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι προέρχονται από την Ουγγαρία. Το ίδιο ισχύει και την σος Ολλανδές, που, την Ολλανδική σάλτσα που είναι σημαντικό αν ε, περιλαμβάνει ένα συγκεκριμένο συστατικό τον κρόκο αυγού ή όχι. Οπότε, ανάλογα με τις ερμηνείες, δημιουργούνται και πολλές προσδοκίες ε, στους επιχειρηματίες των τροφίμων, όπως σημαίνει συνήθως με κάθε νέο κανονισμό. Τώρα, αυτό που περιμένουν οι επιχειρηματίες είναι να είναι σαφής ε, και ξεκάθαρος ο κανονισμός, να μην επιδέχεται διαφορετικές ερμηνείες. Ε, θα πρέπει να περιορίζεται το περιθώριο ερμηνεία των διατάξεων του κανονισμού. Επίσης, οι νέοι κανόνες του εκτελεστικού κανονισμού θα πρέπει να προθεσπίζουν εναρμονισμένου κανόνες ε, για το βασικό κανονισμό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, σε επίπεδο κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, αυτή η τελευταία προσδοκία των επιχειρηματιών ε, προέρχεται από το γεγονός ότι πολλές χώρες ε, θεσπίσουν τις δικές τους διατάξεις ό,τι αφορά την αναφορά της χώρας ή του τόπου προέλευσης. Ε, εδώ μιλούμε για εθνικά συστήματα που δεν είναι γνωστά στους παραγωγούς άλλων χωρών. Ε, επίσης δεν είναι ακόμη γνωστό αν στις ε, συγκεκριμένε διατάξει έγιναν κάποιε αλλαγέ, στα εθνικά συστήματα. Γενικώ ποια είναι η νομική κατάσταση, το νομικό καθεστώς που ισχύει στις διάφορες χώρες. Οπότε δημιουργείται μία αβεβαιότητα για τους επιχειρηματίες. Επίσης, ε, ανακύπτουν ε, ζητήματα όπως η διαφορά στα κριτήρια που χρησιμοποιούνται. για παράδειγμα, οι λιανοπολιτές ή κάποιες αλυσίδες διανομής ε, θα τηρούν τους τοπικούς, τους εθνικούς κανόνες. Δημιουργούνται διαφορετικές προσδοκίες. Επίσης, σε διάφορες αγορές Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ισχύουν εθνικές διατάξεις, δημιουργούνται διαφορετική μεταχείριση μεταξύ εγχώριων παραγωγών και ε, άλλων Τώρα, εμείς θεωρούμε ότι το γεγονό ότι θα εφαρμοστεί εκτελεστικό κανονισμό σε όλε τι χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιφέρει κάποια εναρμόνιση στι κοινοτικέ ρυθμίσει. Επίση, περιλαμβάνει ένα συγκεκριμένο κατάλογο, ε, αρκετά εξαντλητικό σε ό,τι αφορά τα προϊόντα που θα πρέπει να περιέχουν αναφορά προέλευση. Επίση, αναφέρεται περιορισμό σε σχέση με κάποια προϊόντα ως προς την ημερομηνία από την οποία θα, θα ισχύει ο κανονισμός και κυρίως αναφέρει υπάρχει δυνατότητα διαφορετικών ερμηνεών των διατάξεων του κανονισμού λόγω της ε, ασάφειας που περιλαμβάνει ο ορισμός του βασικού συστατικού στον κανονισμό της βάσης, τον 1169. Δεν θα πρέπει λοιπόν να δημιουργούνται διαφορετικές καταστάσεις μεταξύ των επιχειρηματιών λόγω της διαφορετικής ερμηνείας του Τόσο ό,τι αφορά τις ε, προσαρμογές που θα πρέπει να γίνουν στις διαδικασίε διαδικασίες παραγωγής. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τη διαθεσιμότητα κατάλληλων πρώτων σε επαρκείς ποσότητες, την, ποιότητα του... της πρώτης Βέβαια θα πρέπει να δούμε σε τι λεπτομέρειες αναφέρεται ο τόπος προέλευσης. Υπάρχει το θέμα της αποθεματοποίησης. Και υπάρχουν διαφορετικά συστήματα σε ό,τι αφορά το σύστημα αναγνωρισιμότητας ή θα πρέπει να έχουμε καλύτερη προσαρμογή στις διάφορες ε, λήψεις, να έχουμε καλύτερα συστήματα ε, εσωτερικού ελέγχου ποιότητας. Από αυτή την άποψη η παράταση της μεταβατικής περίοδου και η θέση ισχύ από την 1η Απριλίου του 2020 είναι πολύ θετικό για τους επιχειρηματίες για να έχουν μεγαλύτερο διάστημα για να προσαρμοστούν. Σε ό,τι αφορά τους φόβους των επιχειρηματιών, κυρίως είναι ο βασικός φόβος οι διαφορετικές ερμηνείες που μπορεί να δοθούν στο βασικό κανονισμό και που δεν ε, ε, αποτρέπονται από τον εφαρμοστικό κανονισμό. Επίσης, ό,τι αφορά τους κρατικούς ελέγχους των τροφίμων, τους, ε, τις επιθεωρήσεις που θα γίνεται, αλλά και τις υποχρεώσεις των επιθεωρητών. Δυστυχώς υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες που δίνονται στο κανονισμό μεταξύ των επιχειρηματιών και των αρμόδιων φορέων ελέγχου. Οπότε θα έχουμε σημαντικές διαφορές στην διοικητική επιβάρηση ή επιπλέον κόστος λόγω της αλλαγής των ετικετών που θα απαιτηθεί. Όλες αυτές οι διευκρινήσεις είναι πολύ σημαντικές για τους επιχειρηματίες. Είναι πολύ σημαντικό ε, να δοθούν κατευθυντήριες γραμμές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον εκτελεστικό κανονισμό για να απεφευχθούν, όπως είπα, οι αποκλίνουσες ερμηνείες των διατάξεων του εκτελεστικού κανονισμού και του βασικού κανονισμού. Είναι σημαντικό οι καταθεντήρες αυτές γραμμές Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, να περιλαμβάνουν και κάποια παραδείγματα και κάποια, ίσως, ε, κάποιες τυποποιημένες απαντήσεις για τους επιχειρηματίες που θα έχουν πολλές απορίες ως προς την τεχνική εφαρμογή αυτών των διατάξεων. Και τέτοιου είδου κατευθυντήριε γραμμέ θα χρησιμεύσουν ε, και στου επιχειρηματίε αλλά και στου φορεί ε, επιθεώρησης και ελέγχου και θα διευκολύνουν την εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Είμαστε λοιπόν υπέρ ε, του εκτελεστικού κανονισμού, αλλά θα πρέπει να περιοριστεί η βεβαιότητα που δημιουργείται λόγω της δυνατότητας διαφορετικής ερμηνείας. Θα πρέπει να δίνονται πανευρωπαϊκές πληροφορίες σε, σε ό,τι αφορά την σύνθεση των προϊόντων. Ε, χρειάζεται μια πιο εναρμονισμένη προσέγγιση και κατευθυντήριες γραμμές για την πρακτική εφαρμογή του κανονισμού το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ τώρα να πάρει το λόγο ο κ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και εσάς ε, κυρίες και κύριοι αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την οργάνωση της ε, σημερινής για την επισήμανση. Είμαι, λέγομαι Jacobs και είμαι αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Διευθυντής Προφόρησης Καταναλωτών, Διατροφής και Υγείας. Έχουμε 27 κλαδικές ε, ενώσεις, έχουμε 25 εθνικές ομοσπονδίες που αναφέρονται από τη σοκολάτα μέχρι μπύρα και διάφορα άλλα τρόφιμα και ποτά και 21 επιχειρήσεις συνδέσμους. Εάν εξετάσετε τον ε, τομέα παραγωγής και μεταποίησης τροφίμων θα δείτε ότι σε ό,τι αφορά τον κύκλο εργασιών είμαστε από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη και για την απασχόληση το ίδιο και είμαστε ως Ευρώπη και ο μεγαλύτερος εξαγωγίας και είμαστε υπερήφανοι στον κόσμο δηλαδή γι' αυτό. Πολλά από τα τρόφιμα αυτά ε, διοχετεύονται στην ευρωπαϊκή ενία αγορά. Οι πολλοί στην ενία αγορά φτάνουν το 90% του συνολικού κύκλου εργασιών τροφίμων και ποτών. Ε, μεταξύ δε χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αξία είναι περίπου 250 δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, που σημαίνει ότι οι αλυσίδες τροφίμων είναι ενοποιημένες, λειτουργούν διαμεθοριακά και βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλο ε, όγκο εμπορίου πρώτων υλών, είτε πρόκειται για ε, γάλα, ε, κρέμα κλπ. μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών μελών. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, μιας και εορτάζουμε και την 25η επέτειο της ενιαίας αγοράς φέτος. Το 70% τη της παραγωγής των αγροτών μας χρησιμοποιείται ως εισρωές για την μεταποίηση των τροφίμων. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανεξάρτηση μεταξύ γεωργών, αγροτών και μεταποιητών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν εξετάσετε τώρα το νομικό πλαίσιο, πολλά λέχθηκαν ήδη. Υπενθυμίζω ότι εσεί, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και το Συμβούλιο Υπουργών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν ήδη επεκτείνει το νομοθετικό πλαίσιο με τον κανονισμό ε, πληροφόρησης των καταναλωτών, βεβαίω και την επισήμανση, για να μην παραπλανώνται οι καταναλωτές. Υπάρχουν και πολλά εθελοντικά ε, συστήματα και η πρόσφατη ε, νομοθεσία για την ε, επισήμανση της ε, χώρας προέλευσης που είναι ένα πρόσθετο στοιχείο. Συχνά λέγεται ότι η βιομηχανία δεν επιθυμεί τόσο πολύ να παρέχει διαφάνεια για, την, για τους τόπους παραγωγής. Αυτό δεν είναι αληθές όσο όλο και περισσότερο βασίζονται στην αυξανόμενη εμπιστοσύνη των καταναλωτών οι βιομηχανίε. Αλλά για να μπορέσουν να το κάνουν αυτό θα πρέπει να τα αποκρίνονται σε τρία πράγματα. Θα πρέπει να υπάρχει ενδιαφέρον από πλευρά καταναλωτού, θα πρέπει να υπάρχει διάθεση από πλευρά του καταναλωτού να πληρώσει την έξτρα πληροφορία, ακόμα και αν ενδιαφέρεται, και θα πρέπει και ε, λειτουργικά να είναι ε, ε, ε, δυνατόν να εφαρμοστεί, να είναι εφικτό γιατί στις διάφορες αλυσίδες προμήθειας τροφίμων είναι καμιά φορά δύσκολο. Υπάρχουν διάφορα εθελοντικά συστήματα στην αγορά και οι γεωργικές ενδείξεις έχουν αξία της τάξης των 11,5 δισεκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο. Άρα υπάρχει μεγάλη εμπιστοσύνη σε αυτά τα εθελοντικά συστήματα παροχής πληροφοριών για την ε, χώρα προέλευσης, για τα συστήματα μεταποίηση, αλλά και για την υψηλή ποιότητα ε, τροφίμων και μάλιστα η διάθεσή του και στην παγκόσμια αγορά, όπου είμαστε μεγάλος εξαγωγό. Αν δείτε τώρα τα υποχρεωτικά ε, μέτρα, αρχίζουν με τα γαλλικά, που παρουσιάστηκαν ως ένας πειραματισμός με χρονικό περιορισμό. Αν δείτε και τα διάφορα μέτρα θα δείτε ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των μέτρων αυτών όσον αφορά το περιεχόμενο, όσον αφορά τον χρονισμό, όσον αφορά το εάν στο τέλος της ε, πειραματικής περίοδου θα υπάρξει ένα είδος αξιολόγηση στη βάση μιας εκθέσεως. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι πρώτες εκθέσεις θα πρέπει να προκύψουν περί τα τέλη του έτους και θα είναι η χρονική στιγμή όπου θα δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις όχι μόνο στους καταναλωτές αλλά και στις ε, επιχειρήσεις και στο εμπόριο. Αν δούμε τώρα ακριβώς τον αντίκτυπο αυτό θα δούμε ότι ενώ εμφανίζονται ως πειραματικά τα σχέδια αυτά, τα, ε, τα συστήματα αυτά, ο αντίκτυπος της επιχειρήσης ήταν άμεσος Άλλαξαν δηλαδή τις αλυσίδες παραγωγής, τις αλυσίδες μεταφοράς και ούτω καθεξής. Και ενώ υπάρχει μια ρήτρα αμοιβαίας αναγνώρισης, δεν αποκλεί ωστόσο την επανεθνικοποίηση της ε, ε παροχής, δηλαδή τον, ε, για παράδειγμα των σαρκιουτιέφ, των, των αλαντοπιών στη Γαλλία, όπου δεν μπορούν να βασίζονται μονάχα στην γαλλική παραγωγή, παρόλα αυτά προτιμούν τα γαλλικά προϊόντα. Και τώρα αντιμετωπίζουν βέβαια προβλήματα, αντιμετωπίζουν πίεση από μεγάλες αλυσίδες λιανικής πωλήσεως που ζητούν τα προϊόντα αυτά να προέρχονται από τη Γαλλία. Βλέπουμε λοιπόν λιγότερες εισαγωγές, βλέπουμε μείωση κατά 20% εισαγωγών σε ορισμένες περιπτώσεις και 20% βέβαια και κερδοφορίας για τις επιχειρήσεις αυτές. 20% μείωση κερδοφορίας. Και αυτό διότι οι αλλαγές στις πρακτικές, έχει γίνει κατακαιρματισμός έχει γίνει μάλλον διαχωρισμός των, ε, των, των γραμμών παραγωγής αναχώρα και ούτω καθεξής. Και ας μην λησμονούμε και τις αναποτελεσματικότητες που θα προκύψουν. Βλέπουμε και αντίκτυπο στο ένδο ενωσιακό εμπόριο. Και εκ του λόγου αυτού αντιμετωπίζουμε υψηλότερες τιμές πρώτων υλών που μπορούν να καταλήξουν και σε υψηλότερε τιμέ καταναλωτού. Και νομίζω ότι έχει γίνει και μια συζήτηση ήδη, δηλαδή τη τιμή καταναλωτού την ορίζει ο λιανικός έμπορος και όχι ο αρχικός παραγωγός. Επομένω, δηλαδή αυτά μπορούν να καταλήξουν σε υψηλότερες τιμές καταναλωτών. Και εν πάση περιπτώσει αυξάνεται επίσης το σύστημα. Ο αντίκτυπος είναι μεγαλύτερος για μικρές επιχειρήσεις. Για αυτές που είναι σε μεθοριακές περιοχές καθώς και για επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ποικίλε πηγές για τις πρώτες ύλε τους. Και είχε γίνει έκθεση προετών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έδινε μια πρώτη γεύση εφόσον επιλέγεται ε, για παράδειγμα κρέας από ε, μία χώρα μπορεί να φτάσουν μέχρι και τα 50% αύξησης του κόστους. Υπάρχει λοιπόν αρνητικός αντίκτυπος κάποτε θεωρούταν θεωρητικός. Τώρα βλέπουμε όμως το πραγματικό αντίκτυπο στην αγορά και βλέπουμε για παράδειγμα σημαντική μείωση των βελγικών εξαγωγών ε, γάλακτος στην ε, Γαλλία μετά από την ε, πρόσφατη γαλλική νομοθεσία. 17,7% μείωση των βελγικών εξαγωγών γάλακτος στη Γαλλία τις τρεις πρώτους μήνες. Δεν είναι κάτι λοιπόν που μπορεί να το πάρει κανείς αψήφιστα. Μίλησα για το γάλα, αλλά ακόμα και η σκόνη γάλακτος, οι εξαγωγές ε, γάλακτος σε σκόνη προς την Γαλλία έχουν εξαφανιστεί. Βλέπετε λοιπόν ποιες είναι οι αρνητικές επιπτώσεις αυτής της εθνικής υποχρεωτικής ε, προσέγγισης που μπορεί να έχει δηλαδή στο εμπόριο και στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Το ίδιο ισχύει για τη Γερμανία. Εξαγωγές δηλαδή Γερμανίας προς Γαλλία και μπορώ να θυμίσω και παραδείγματα από τη όπου οι εξαγωγέ κρέατος από τη Σουηδία στη Γαλλία έχουν μειωθεί κατά 30%. Βλέπουμε λοιπόν τι πρώτε πρώτες επιπτώσεις στην πραγματική ζωή της αγοράς. Έχουμε τώρα και άλλες ανησυχίε νομικές, διαδικαστικέ κλπ. Και πρώτα ο κανονισμός ΦΙΚ που λέει ότι οι χώρες θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες διασύνδεσης μεταξύ των διαφόρων φάσεων παραγωγής κλπ. Καμιά χώρα δεν το έχει κάνει αυτό. Θα πρέπει ωστόσο να αποδείξουν επίση ότι υπάρχει ενδιαφέρον του καταναλωτού. Μιλούμε για, για, γνήσιο ε, ενδιαφέρον του καταναλωτού ή μιλούμε για άλλους στόχους. Υπάρχει για παράδειγμα ισπανικό διάταγμα το οποίο λέει ρητά ότι λαμβάνουν το μέτρο αυτό για λόγους προστατευτισμού. Είναι λοιπόν πραγματικά αυτό ο σκοπό μήπω των μέτρων. Επίση πρέπει να εξετάσουμε και τον σεβασμό του κράτους δικαίου. Βλέπουμε χώρες όπως η Ιταλία αλλά και η Ρουμανία που έχουν εγκρίνει νομοθεσία χωρίς να, κοινοποιήσουν, να την κοινοποιήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το οποίο βεβαίως δεν είναι σύμμορφο με τις διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχει και το διεθνές στοιχείο, διότι οι διεθνείς εμπορικοί εταίροι μας δεν εκφράζουν ιδιαίτερη ικανοποίηση. Ο Καναδάς την προηγούμενη εβδομάδα ε, δήλωσε, ανακοίνωσε ότι σκέπτεται να προσφύγει στη, στον ΠΟΕ, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Η Ιταλία, η Ιταλία επίσης για θέματα ζυμαρικών. Αλλά η σχετική νομοθεσία που εγκρίνουν οι χώρες μέλη πρέπει να κοινοποιείται και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Ούτε για μας είναι εύκολο να έχουμε συνολική επισκόπηση που βρίσκονται αυτές οι, ευρωπαϊκές οι εθνικές νομοθεσίες, τα διάφορα διατάγματα δηλαδή. Ανέφερα ήδη τις μελέτες αντικτύπου που φαίνεται να έχουν αγνοηθεί σε ορισμένε από τι περιπτώσει αυτέ και φαίνεται οι ίδιε οι μέρε αντικτύπου να έχουν αγνοήσει το στοιχείο του κόστου και τελικώ και στον καταναλωτή και την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών αλυσίδων προμηθειάς τροφίμων. Έχουμε τώρα βέβαια και την επισήμανση της προέλευσης των βασικών συστατικών. Θα συμφωνήσω με τη συνάδελφό μου, χωρίς να θέλω να μακρηγορήσω, ότι θα ήταν σωστό να υπάρξει μια ενιαία προσέγγιση, αλλά αναμένουμε αυτό να σημάνει και το τέλος των εθνικών μέτρων. Η συνύπαρξη εθνικών και κοινοτικών μέτρων είναι κάτι το μη επιθυμητό και βεβαίως είναι και ανέφικτο για τις επιχειρήσεις και κάποιες χώρες οι οποίες έχουν εγκρίνει εθνικά διατάγματα έχουν αναφέρει ρητά ότι θα διακόψουν τα εθνικά, την ισχύ των εθνικών διαταγμάτων εάν τα μέτρα αυτά για την επισήμανση δηλαδή των βασικών συστατικών εγκριθεί. Τώρα λοιπόν αυτό έχει αρχίσει, το νομοθέτημα έχει αρχίσει να ισχύει και αναμένουμε λοιπόν επομένως τα σχετικά μέτρα να εξαφανιστούν. Τέλος, η έλλειψη διαφάνειας που πρέπει επίσης να αντιμετωπιστεί. Επεξεργαζόμαστε έναν εναρμονισμένο ε, κώδικα για την βιομηχανία, για την εφαρμογή των σχετικών νομοθεσιών. Εν τέλει, θα ήθελα να τονίσω ότι οι αλυσίδες προμήθειας τροφίμων δεν πάβουν να ισχύουν από τα σύνορα μιας χώρα και πέρα. Καμία χώρα μέλο τη Ένωση δεν είναι σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα. Όλες εξαρτώνται από άλλε. Οι supply chains έχουν δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αποτελεσματικές, αποδοτικές να αποφεύγουν την σπατάληση τροφίμων όσο αυτό είναι δυνατό, να στηρίζουν την βιωσιμότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων σε ολόκληρη τη διάρκεια του έτους, αν θέλουμε να ακολουθήσουμε την οδό των εθνικών ρυθμίσεων, εθνικών μέτρων, θα χάσουμε το πιο σημαντικό στοιχείο της Ένωσης μας, που είναι η ενιαία αγορά. Εν τέλει, ουδής κερδίζει από αυτές τις εθνικές προσεγγίσεις. Όλοι τελικώ θα είμαστε χαμένοι και τελικώ δεν θα κερδίσει κανείς. Αυτό που έχουμε τώρα είναι ένα πλήρες σύνολο κανόνων νομοθεσίας που αποτρέπουν την παραπλάνηση των καταναλωτών. Κάθε φορά που υπάρχει ενδιαφέρον, κάθε φορά που υπάρχει επιθυμία ο καταναλωτής να πληρώσει κάτι παραπάνω και αυτό είναι και εφικτό, έχει καλός. Τότε ε, πράγματι ε, βιομηχανίες, οι επιχειρηματίες, ας το πράξουν. Αλλά ας μείνουμε σε εθελοντική βάση αντί να προσπαθούμε να βγάλουμε το μάτι των δε. Ευχαριστώ πολύ. ο κύριος Κάρας. Έχετε λόγο. Ο κύριος Κάρα. Καλημέρα σε όλους. Χρειάζομαι τις διαφάνειες. Καλημέρα σε όλους. ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είμαι ο Παύλο Καρά, πρόεδρο ε, του Εθνικού Φορέα Ρίζη. Ε, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μα δίνετε σήμερα να μιλήσουμε για το Ιταλικό Ρίζη και το Ευρωπαϊκό Ρίζη στα πλαίσια της ετικετοθεσίας. Εν συντομία, η Nationale Ρίζη είναι ένας φορέας δημόσιος οικονομικός υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Δασοκομείας και Γεωργίας Ιταλίας. Αποστολή μας είναι να υπαρασπιστούμε την εθνική παραγωγή του προϊόντος ταυτόχρονα μέσω του κέντρου ερευνών να βρίσκουμε λύσεις. Λύσεις για καλλιέργεια ρυζιού με βιώσιμο τρόπο και Βρισκόμαστε σε αυτή την αλυσίδα και το Διοικητικό μας Συμβούλιο αποτελείται από παραγωγούς και μεταποιητές και ο υποφαινόμενος είναι παραγωγός, είναι ριζοπαραγωγός στην Ιταλία. Η Ιταλία είναι πρώτη χώρα σε παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 52,20% παραγωγή. Μετά ακολουθεί η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Ουγγαρία αλλά αντιπροσωπεύει μόνο το 0,2% της παγκόσμιας παραγωγής παρόλα αυτά η Ιταλική παραγωγή. Ένα από τα χαρακτηριστικά της ριζοκαλλιέργειας Ιταλικής είναι ότι εν ονόματι των διαφόρων ποικιλιών, καρναρόλι, αρμπόριο, βιαλόνι, νάνος, αυτά τα προϊόντα έχουν γίνει εμπορικά σήματα θα έλεγα, ονομασίες προϊόντων. Και υπενθυμίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, αναγνώρισε την ευρωπαϊκή ριζοκαλλιέργεια και θεωρείται ένα δημόσιο αγαθό από πλευράς περιβαλλοντικής. Το ρύζι που καλλιεργείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα προϊόν βιώσιμο από πλευράς περιβαλλοντικής και παρέχει εγγυήσει στον καταναλωτή όσον αφορά την υγεία. Αυτά τα χαριστικά δεν τα βλέπουμε στο ρύζι εισαγωγής πάντα. Βλέποντας λοιπόν του συναγερμούς, τις ειδοποίησεις της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασφαλείας των Τροφίμων, πολύ σημαντικά βλέπουμε εισαγωγή ρυζιού βασμάτη, ε, περιλαμβάνει ίχνη ε, παρασιτοκτόνου όπως το καρπενταντζίμ, το οποίο είναι ένα προϊόν που απαγορεύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, το 2006 ο τομέας ο Ιταλικός του ρυζιού και Ευρωπαϊκός αντιμετώπιζε πρόβλημα στον αφορά από τις Ηνωμένε Πολιτείε που ε, είχε ίχνη προϊόντων γενετικά τροποποιημένων. Η απάντηση της Ιταλίας αυτή την εποχή ήταν να εθελοντικά να εφαρμόζουμε ένα σήμα που το βλέπετε εδώ. Βλέπετε κόκκους, πράσινους, λευκούς και ρυθρούς και με τη σφαγίδα ιταλικό ρύζι που διαχειριζόταν η National Rizzi και αυτό το σήμα έχει καταχωρηθεί διεθνώ, που καθορίζει την προέλευση, τη φύση και την ποιότητα του Ιταλικού ε, ρυζιού που πωλείται από του Ιταλού εμπορευμα... Ε, ε, εμπόρου. Λοιπόν, το Ιταλικό ρύζι, ρύζο Ιταλιάνο, αυτό το σήμα είναι μια καλή απάντηση για να βρούμε μια απάντηση στα προϊόντα με κατάλοιπα γενετικών τροποποιημένων οργανισμών. Λοιπόν, ο τίτλο είναι Το Ευρωπαϊκό Ρύζι τη παρουσιάσεω μου. Το Ιταλικό ρύζι δεν είναι κομμόντι, δεν είναι βασικό προϊόν, διότι κατά κάποιο τρόπο το Ιταλικό ρύζι έχει καθορισμένε ποικιλίε, ποικιλίε που χρησιμοποιούνται για υποετοιμασία διαφόρων εδεσμάτων. Ένα, μια άλλη μάρκα, ένα άλλο μπραντ είναι αυτό που συνδέεται με το ριζότο, ε, μια τυπική συνταγή, αλλά και συνταγές που αφορούν ε, σημαντικά άλλα φαγητά το ρύζι που καλλιεργείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά τα χρόνια έχει προβλήματα από τις εισαγωγές με μηδενικό τέλος. Τα τελευταία δέκα χρόνια οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 50% και τώρα το μισό της κατανάλωσης ρυζιού στην Ευρώπη ε, καλύπτεται από εισαγόμενο ρύζι. Το 25% του ρυζιού που εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση προέρχεται από χώρες στις οποίες για τους λόγους που προανέφερα διαφύλαξη του περιβάλλοντος, ο σεβασμός των ε, πολιτικών δικαιωμάτων δεν εφαρμόζονται όπως είναι η Καμπότζη, Φερρυπίν, μια από τις χώρες. Και διαβάστε το έγγραφο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε στην, στην, ε, μέσω της εταιρείας Development Solutions και εκεί εστιάζεται το έγγραφο επί της ζάχαρης και του ρυζιού σχετικά με την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην παραγωγή των προϊόντων. 23 Ιανουαρίου αυτού του έτους στις Βρυξέλλες η International Ρίζη διοργάνωσε ένα δεύτερο συμπόσιο με θέμα το ευρωπαϊκό ρύζι και εκεί στις συζητήσεις διεφάνει και η ανάγκη να, γίνονται, να γίνεται σεβαστή η αμοιβαιότητα για θέματα κοινωνικά, το δικαίωμα εργασίας και για θέματα περιβάλλοντος. Και μετά έχει αντιμετωπίσει το φαινόμενο του Italian Sounding. Το μιμούνται. Βλέπετε στη φωτογραφία, το ιταλικό ρύζι το μιμούνται. Αρμπόριο ράις, συσκευασία αρμπόριο ράις για ριζότο. Στην πραγματικότητα, αυτό το, στο αυτό το κουτί δεν υπάρχει ιταλική ποικιλία. Όπως σας έλεγα, υπενθυμίζει την αρμπόριο, μια ποικιλία που είναι και εμπορικό σήμα, αλλά το περιεχόμενο είναι ένα ρύζι που δεν χρησιμοποιηθεί για ριζότο, αλλά όπως βλέπετε και στη φωτογραφία ε, χρησιμοποιείται σαν ε, προϊόν για συνοδευτικό στο ρύζι. Ε, λοιπόν, ίσως απομακρύνθηκα κάπως για να φτάσω προς το τέλος της παρεμβάσεώς μου. Θέλω να σας πω ότι ο ριζοπαραγωγή Ιταλή, στη μεγάλη τους πλειοψηφία είναι υπέρ όχι μόνο η τοκετοθεσία που θα αναφέρει την προέλευση, αλλά αυτή η τοκετοθεσία να είναι υποχρεωτική και ένα μικρό τμήμα των παραγωγών ε, θεωρούν ότι δεν θα λύσει όλα τα προβλήματα του τομέα αυτή τη δικαιοθεσία, αλλά αυτό που διακρίνει τους Ιταλούς παραγωγούς και τολμώ να πω τους Ευρωπαίους παραγωγούς από τους μεταποιητές, από τους rice millers, αυτοί που ε, αυτοί προτιμούν θελοντική εφαρμογή της δικαιοθεσίας, αυτοί που εξεργάζονται το ρύζι, οι rice millers. Ε, ε, εμείς ε, θέλουμε να αναφέρετε το Made in Italy, Italian Made. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε και εμείς κύριε Καρά. Και τώρα κύριε Νικολακοπούλου, εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής Διτσισάντε. Thank you very much, uh, Madam. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά την Επιτροπή για την πρόσκληση αυτήν την ανταλλαγή απόψεων με θέμα τον εκτελεστικό κανονισμό για την επισήμανση της προέλευσης και μάλιστα τόσο γρήγορα μέσω μετά την έγκριση αυτή του, αυτού του εκτελεστικού κανονισμού. Ακούσαμε πολλά για τον εκτελεστικό κανονισμό, τον αντίκτυπο που έχει τις συνέπειες του, κατά πόσο ικανοποιεί τις προσδοκίες του καταναλωτή, στην απέτηση του για διαφάνεια και επίσης ε, ακούσαμε την... τα αιτήματα από πολλές πλευρές στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προβλέψουμε υποχρεωτική αναφορά της προέλευσης. Και μάλιστα ο εκτελεστικός κανονισμός αποτελεί το αποτέλεσμα εντατικών συζητήσεων που ξεκίνησε και από την προηγούμενη θητεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μάλιστα ο κανονισμός, όταν εγκριθήκε ο κανονισμός για την, την νομοθεσία των τροφίμων το θέμα της αναφοράς προέλευσης ήταν από τα πιο φλέγοντα και επίμαχα ζητήματα, ζητήματα που δίχασε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη τελικά καταλήξαμε σε μια συμβαστική λύση προκειμένου να ενισχύσουμε τους κοινοτικούς κανόνες και για πρώτη φορά έχουμε και την, τον ορισμό της ε, επισήμανσης ε, προέλευσης ε, που αναφέρεται στο κανονισμό και το τελωνιακό και που υποχρε... θεσπίζει υποχρεωτική αναφορά της προέλευσης για κάποια ε, προϊόντα όπως κρέας. Ε, συζητήθηκε το θέμα της υποχρεωτικής αναφοράς ε, της προέλευσης και για άλλες κατηγορίες προϊόντων, αλλά δεν επετεύχθη συμφωνία και υποσχεθήκαμε να εκπονήσουμε διάφορες μελέτες για τα για το κατά πόσο για συστατικά κρέατος, γάλα, συστατικά γάλακτος και το κύριο συστατικό μεταποιημένων, επεξεργασμένων προϊόντων θα χρειαζόταν υποχρεωτική αναφορά προέλευσης. Το αποτέλεσμα όλων των μελετών έδειξε ε, θετική απήχηση της διάταξης για τους καταναλωτές και επίσης διαπιστώσαμε θετικές επιπτώσεις ό,τι αφορά την πρόθεση της εχώριας παραγωγής ε, των Ευρωπαίων αγροτών, κάτι που τους εξυπηρετεί. Αλλά διαπιστώθηκαν κάποιες αρνητικές συνέπειες ό,τι αφορά την εσωτερική αγορά και κυρίως ε, αύξηση του κόστους και ε, ε, διοικητική, αύξηση της διοικητικής επιβάρησης των επιχειρηματιών τροφίμων. Και μάλιστα καταλήξαμε για υποχρεωτική αναφορά, σε υποχρεωτική αναφορά της προέλευσης για συγκεκριμένα προϊόντα και εθελοντική για άλλα προϊόντα. Κρίναμε ότι αυτή είναι η πιο ισορροπημένη προσέγγιση για να εξασφαλίσουμε διαφάνεια στην αγορά. Τώρα, για ένα άλλο θέμα που δεν είναι η υποχρεωτική αναφορά προέλευσης ε, για όλα τα τρόφιμα, είχαμε και έναν άλλο κανόνα που στόχο είχε να εξασφαλίσει ότι όταν η αναφορά προέλευσης χρησιμοποιείται ως ε, μέσο για την πρόθεση, και τη διαφήμιση προϊόντων στην εσωτερική αγορά, να μην παραπλανεί τους καταναλωτές, να μην τους παραπληροφορεί και να περιέχει ακριβείς πληροφορίες. Γι' αυτό ο κανονισμός για, την, για τις πληροφορίες και το τρόφιμα προβλέπει την απέτηση σε περίπτωση ε, επισήμασης προέλευσης που δίνεται εθελοντικά να αναφέρεται και η προέλευση του κυρίου συστατικού αν αυτή είναι διαφορετική από την προέλευση του τελικού τροφίμου ή να επισημαίνεται αυτή η διαφορά χωρίς ε, να δίνει ακριβείς πληροφορίες να αναφέρει τουλάχιστον ότι η προέλευση του βασικού συστατικού δεν συμπίπτει με την προέλευση του τελικού τροφίμου. Και αυτός ο εκτελεστικός κανονισμός ε, έπρεπε κανονικά να έχει εγκριθεί ήδη από το 2013 προκειμένου να ισχύσει από το 2014 μαζί με τον κανονισμό ε, για τις πληροφορίες για τα τρόφιμα. Τελικά εγκρίθηκε μόλις πρόσφατα, πριν από λίγες μέρες, με σημαντική καθυστέρηση δηλαδή, λόγω ε, της διαμάχης που προέκυψε και της ε, διάστασης απόψεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Κρατών Μελών και της ανάγκης διαπραγματεύσεων προκειμένου να βρεθεί συμβαστική λύση. Αυτό ο εκτελεστικός κανονισμός θα αρχίσει να εφαρμόζεται από το 2020, οπότε θα μπορέσουν οι υπεύθυνοι επιχειρήσει τροφίμων να, ε, να καταφέρουν να προσαρμοστούν ε, σε αυτή τη μεταβατική περίοδο και επίσης αναφέρονται κάποιες γεωγραφικέ περιοχέ για τις οποίες αναφέρεται η προέλευση και επίσης προβλέπει και κατάλογο ε, των τρόπων παρουσίας αυτών των πληροφοριών, ώστε οι πληροφορίες ε, σχετικές να είναι όρατες, ευανάγνωστες και να προστίθεται στην επισήμανση της προέλευσης του τελικού προϊόντος, του τελικού τροφίμου. Παρά βέβαια την, έγκριση του εφαρμοστικού κανονισμού, του εκτελεστικού κανονισμού, έχουμε και πολλά εθνικά συστήματα. Εφτά κράτη-μέλη έχουν ε, κοινοποιήσει και εγκρίνει εθνικούς κανόνες για την υποχρεωτική επισήμαση ε, προέλευσης ε, για ε, το κρέας, ε, για προϊόντα που περιέχουν κρέας, για το γάλα και προϊόντα που περιέχουν γάλα. Και μάλιστα τα μέτρα αυτά έχουν πειραματικό χαρακτήρα, είναι χρονικά οριοθετημένα και περιορισμένα. Τα περισσότερα τέτοια εθνικά συστήματα θα εκπνεύσουν το αργότερο το 2019 και τα κράτη-μέλη έχουν αναλάβει τη δέσμευση να ε, παράσχουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μία έκθεση που θα εξηγεί τον αντίκτυπο της συνέπειας αυτών των εθνικών κανόνων και στους καταναλωτές αλλά και στο εμπόριο γενικά και στην εσωτερική αγορά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη στιγμή που θα λάβει τις σχετικές εκθέσεις των κρατών μελών με την αξιολόγηση των εθνικών συστημάτων θα τις μελετήσει πολύ διεξοδικά και θα δει ποιες είναι, τα αποτελέσματά τους και τι ε, επίπτωση θα έχουν στις μελλοντικές στρατηγικές και πολιτικές οι νομοθετικές προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα εθνικά πάντως μέτρα θα εκπνεύσουν κάποια στιγμή και δεν προβλέπεται αυτόματη ανανέωσή τους. Αν κάποια χώρα μέλος θέλει να συνεχίσει να παρατείνει την εφαρμογή αυτών των μέτρων, θα χρειαστεί να υποβάλει νέα κοινοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι αλήθεια ότι δεν το έχουν κάνει αυτό όλα τα κράτη-μέλη. Γιατί η εξέλιξη αυτή δείχνει ακριβώς ε, την πορεία των συζητήσεων που είχαμε τα τελευταία χρόνια. Τα κράτη-μέλη που ήταν υπέρ των υποχρεωτικών διατάξεων για την επισήμανση της προέλευσης ε, απογοητεύτηκαν από τα ε, αποτελέσματα της έκθεσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής και απογοητεύτηκαν από τις μεγάλες καθυστερήσει ό,τι αφορά την έγκριση του εκτελεστικού κανονισμού. Γι' αυτό και προχώρησαν στην ε, θέσπιση εθνικών μέτρων. Αλλά ήταν λίγα τα κράτη-μέλη που έκαναν κάτι τέτοιο. Η πλειοψηφία δεν υιοθέτησε εθνικά συστήματα. Αυτά. Θα ήθελα πάντως να προσθέσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη ανέλαβε τη δέσμευση να συνεργαστεί με τα κράτη-μέλη προκειμένου να δώσει τις απαραίτητες διευκρινήσεις ε, για να αποφευθούν παρερμηνίες του εκτελεστικού κανονισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα μέλη του πάνελ. Α ακούσουμε τώρα ερωτήσεις και να δοθούν και απαντήσεις ερωτήσεις. Πάμε σε αυτό το τμήμα της συζήτηση. Έχω κάποια ονόματα εδώ. Αν κάποιος άλλος θέλει να λάβει χώρα στη συζήτηση, α μου το δηλώσει. Ο κ. Έρντος είναι ο πρώτος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και εσείς, κυρίες και κύριοι εμπειρονόμονες, επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω ότι 1η Μαρτίου εγκρίθηκε ο κανονισμό για το μέλι με υποστήριξη 4 πέμπτων των Ευρωβουλευτών και αναμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τις χώρες μέλη να εξασφαλίσουν την βάση για υψηλής ποιότητας εμπόριο μελιού και να αντιμετωπίσουν ιεσδήποτε απόπειρες απατών που μπορεί να προέλθουν από έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν έμποροι οι οποίοι αναμειγνύουν το μέλι και έτσι εξαπατούν τον καταναλωτή. Φαίνεται πως η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται χρησιμοποιούνται προϊόντα, ε, ακόμα και προϊόντα ρητίνης τα οποία αναμειγνύονται με ευρωπαϊκά μέλια, ορισμένα από αυτά από την Κίνα, τα οποία αναμειγνύονται με ευρωπαϊκά μέλια και φτάνει τελικώς ουγγρικό μέλι ακακίας να είναι φθηνότερο στην αγορά από ότι ακόμη και απλό μέλι. Αυτό θα είναι καταστροφή για τον τομέα. Πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος αυτός. Πώς είναι δυνατόν να προστατευθούν οι παραγωγοί. Πώς είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί ότι οι παραγωγοί θα προσφέρουν πραγματικά ευρωπαϊκό μέλη στις ευρωπαϊκές αγορές. Αρκούν οι ρυθμίσεις σε εθελοντική βάση. Τι πρέπει να γίνει για να αποφύγουμε την ε, προσφορά στο, στην ευρωπαϊκή αγορά αυτών των νοθευμένων προϊόντων μελιού. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Εύανς, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους καλεσμένους μας εμπειρογνώμονες. Σε ό,τι αφορά το ρύζι, την ε, περίπτωση που μας παρουσίασε ο κύριος Καρά. Και εμάς μας προβληματίζει ιδιαίτερα στο θέμα του ρυζιού και με τον κύριο Δεκάστρο στείλαμε επιστολή στην Επιτροπή Wallstrom και είχαμε και κοινοβουλευτική ερώτηση. Μία το Φεβρουάριο με απάντηση ε, τον Απρίλιο, δεύτερη επιστολή είχε ημερομηνία 31 Μαΐου την περασμένη εβδομάδα και καταφέραμε να εκβεύσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ε, την ε, επιβεβαίωση μας έδωσε εδώ και πάρα πολύ καιρό η Κόπα Κοζέκα και το μαγετορίζει. Ε, έχουμε την περίπτωση της συμφωνίας με την Καμπότζη, με τη Μερκοσούρ, ε, ο, ο, το μέσο ριζοκαλλιέργειας επλήγει ιδιαίτερα από τη συμφωνία όλα με εξαίρεση τα όπλα και ιδιαίτερα αυτή η συμφωνία ήταν πολύ επιβαρυντική για τους ε, οριζοκαλλιεργητές. Θεωρείτε ότι η επισήμαση πρόελευση στο ιταλικό προϊόν ή το ισπανικό προϊόν made in Italy, made in Spain είναι αρκετή διάταξη. Μήπως θα έπρεπε ταυτόχρονα να έχουμε και ένα ειδικό πρόγραμμα στα πλαίσια του κανονισμού προώθησης, γιατί αν δεν καταφέρουμε να προωθήσουμε τα προϊόντα μας ώστε να γνωρίζει ο καταναλωτής την προέλευση του ρυζιού, προς τι το σήμα ιταλικό προϊόν, το made in Italy, αν ε, δεν έχουμε δώσει κίνητρα στον καταναλωτή να αγοράσει αυτό το τελικό ρύζι. Και τέλος θεωρείτε ότι προλαβαίνουμε να σώσουμε τον κλάδο του ρυζιού γιατί στην Ισπανία για παράδειγμα έχει περιθωριοποιηθεί τελείως ε, η οριζοκαλλιέργεια ακόμη και στη Βαλένθια που ήταν κατεξοχή οριζοπαραγωγός περιοχή. Και περιοχές όπως η Καταλανία, η Μούρσια, η Αντα... Ανταλουσία που παλιά είχαν ε, ένα θαλερό κλάδο ρυζιού έχουν πια καταστραφεί και είναι αδύνατο να τον επαναφέρουμε και να τον αποκαταστήσουμε. Ο κύριος Αντρίε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν εκπλήσωμε από την απάντηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συνηθίζουμε μετά από τι διάφορες συνεδριάσεις και τους μήνες που περνάνε αλλά εκπλήσωμε. Συγγνώμη από αυτή την έλλειψη συνέπειας θα έλεγα. Το λέω μα είχαμε εμπειρία ε, που παραμένει σήμερα. Λοιπόν, δεν λάβατε καθόλου υπόψη την άποψη της, ε, του Ευρωκοινοβουλίου σε αυτά που κάνατε. Το να μην γίνει αξιολόγηση μετά από 8 διαφορετικά πειράματα που έγινε στην Ευρώπη, θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι που με εκπλήσει δεν θα πρέπει να, να παραμείνουμε... Να... Κοιτάξτε, η τεχνολογία προχωρά γρήγορα, δεν πρέπει να μείνουμε πίσω. Λοιπόν, να μην αποξηρανθούμε σαν φυτά. Λοιπόν, η τεχνολογία προχωρεί πάρα πολύ γρήγορα. Θα πρέπει να προσέξουμε και θα πρέπει κάτι να, σε κάτι να χρησιμεύει τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγγνώμη που το λέω ομά. Είναι κατεπίγουσα η ανάγκη. Οι καταναλωτέ σήμερα είναι πάρα πολύ απαιτητική όσον αφορά την προέλευση. Το είπατε γίνανε κάποια πειράματα, αλλά όχι μόνο για την προέλευση, για τη σύνθεση των τροφίμων. Ε, ε, λοιπόν, ε, υπάρχει ενδιαφέρον για την ανθρώπινη υγεία. Υπάρχουν αναδυόμενες ασθένειες λόγω καρκινογόνων, προβλήματος με το πάγκρεας, παχυσαρκίες κλπ. κλπ. Κάνουμε διάφορες ακροάσεις και ακούμε όλο και περισσότερα προβλήματα. Λοιπόν, είναι κατεπίγουσα η ανάγκη επιτάχυνση των διαδικασιών. Αυτό θέλω να πω, κυρία Πρόεδρε. Λυπούμε. Αλλά νομίζω ότι σήμερα πραγματικά να προχωρήσουμε. Διότι γίνονται κάποια πειράματα Λοιπόν, θα πρέπει να δούμε ότι είναι κατά επίγουση ανάγκη. Αν δούμε ότι ε, περιμένουμε να γίνει αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 8 πειραμάτων, περιμένουμε και όλα αυτά, φοβάμαι ότι θα προχωρήσουν πιο γρήγορα απαιτήσει των πολιτών και οι χρόνοι. Και εμεί χρονοτριβούμε. Μπορούμε... Λοιπόν, πρέπει να προχωρήσουμε πιο γρήγορα. Χρειάζεται επιτάχυνση. Δεν είναι θέμα ίσονο σημασία καθόλου. Συγγνώμη για αυτή την παρέμβαση, κυρία Πρόεδρε, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να ξυπνήσουμε. Διότι αυτά τα θέματα της προέλευσης δεν είναι μόνο θέμα προέλευσης. Το θέμα των τροφίμων, της πληροφόρησης των καταναλωτών, των 500 εκατομμυρίων καταναλωτών που εκπροσωπούμε. Και πρέπει να σας πούμε, κύριε εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι θέμα πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει όλη η διαδικασία να επιταχυνθεί. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ντόλφμαν έχει το λόγο. Και εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στο ρύζι και να συνεχίσω σε αυτά που είπε η συνάδελφος Έραντς. Σίγουρα ότι αναφορά της προέλευσης μπορεί να συμβάλλει στη λύση. Θεμελιώδες πρόβλημα όμως είναι ότι εμείς κατά την άποψή μου ε, προερχόμαστε από μια χώρα ε, όπου ε, στι διαπραγματεύσει χώρα προέλευση αυτού του προϊόντο, τα everything but arms, στι διαπραγματεύσει. Δεν λαμβάνει υπόψη κάποιε συνθήκε που επικρατούν εκεί. Δεν είναι δημοκρατική χώρα η Καμπότζη, η Φερρυπίν. Ακόμα χειρότερα, και χειρότερο για μας και καλύτερο για αυτούς είναι μια χώρα όπου δεν έχει πλέον δεν μπορεί να παραμείνει στα πλαίσια του everything but arms, τα πάντα εκτός από όπλα, στα πλαίσια της συμφωνίας. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν ποια είναι η κατάσταση σε μια χώρα επί τόπου και να περιμένουμε χρόνια και χρόνια μέχρι να αλλάξουν οι τελωνιακές προτιμήσεις. Εγώ πάντα προάσπιζα το everything but arms, αλλά κάποιες χώρες όπως είναι η Καμπότζη και άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας είναι πραγματικό πρόβλημα για το ρύζι και θα πρέπει να βλέπουμε ποια κατάσταση επικρατεί εκεί. Το, το, για το μηδενικό τέλος που ισχύει μόνο για το ρύζι αλλά και για άλλα προϊόντα και δεν έχει λόγο ύπαρξης πλέον στα πλαίσια αυτών των συμφωνιών Everything But Arms. Ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να μιλήσει η κυρία Κάντεμπαχ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ για τις ε, τοποθετήσεις και μπορώ νομίζω να συνεχίσω αμέσως μετά τα όσα είπε ο Ντόρφμαν. Πρέπει να εξετάσουμε όλο μαζί αυτό το project της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συχνά συζητούμε ξεχωριστά πράγματα, σε σιλό αγροτική πολιτική, πολιτική υγείας, ε, ε, ενιαία αγορά και ούτω καθεξής. Τα ζητήματα όμως που συζητούμε σήμερα είναι τέτοια που δεν μπορούν να χωριστούν, να μπουν με το ζόρι σε αυτά τα σιλό. Ιδίω η επισήμανση των προϊόντων μπορεί να συμβάλλει και χωρίς να θέλουμε να είμαστε προστατευτικοί. Μπορούμε όμως α, να δώσουμε την δυνατότητα στον καταναλωτή να αποφασίσει, δηλαδή να λάβει μια απόφαση βασισμένη σε γνώση. Να γνωρίζει ότι το προϊόν προέρχεται από την τάδε περιφέρεια και θέλω να συμβάλλω. Ας πούμε και για την αποφυγή της επιβάρυνσης του κλίματος, ώστε να είναι όσο το δυνατόν συντομότερες οι οδοί μεταφοράς. Για παράδειγμα, για να διατηρηθεί απασχόληση στη συγκεκριμένη περιφέρεια, για να ε, υπάρξει μια ποιότητα ε, ζωής. Επομένως, μπορεί να λαμβάνει στοχευμένα συγκεκριμένες αποφάσεις μέσα σε μια επιθυμία να υποστηρίξει μια συγκεκριμένη περιφέρεια. Ω καταναλώτρια μπορώ να το πράξω αυτό μόνο αν γνωρίζω από πού προέρχεται το προϊόν. Αν θέλουμε λοιπόν πολιτική συνοχή, πολιτική κλίματο, πολιτική περιβάλλοντο, αλλά τελικά και εμπορική πολιτική, τότε χρειαζόμαστε τι επισημάνσει αυτέ. Διότι αλλιώ ω καταναλώτρια δεν μπορώ να λάβω τι σχετικέ αποφάσει. Και αυτό νομίζω ότι δεν έχει σχέση με οποιοδήποτε προστατευτισμό. Έχει σχέση με το γεγονό ότι θέλω συνειδητά να μπορώ να πω ω καταναλώτρια θέλω να διατηρήσω σε ζωή μια περιφέρεια, μια συγκεκριμένη περιφέρεια. Θέλω προϊόντα από την περιφέρεια αυτή, θέλω να είναι μικρέ οι αποστάσει που διανύουν τα προϊόντα μέχρι να φτάσουν σε μένα. Ε, νομίζω ότι χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια εθελοντική επισήμανση. Χρειαζόμαστε μια απόφαση που να προσφέρει τη δυνατότητα αυτή τη καταναλωτή και όχι μόνο για το ρύζι, γενικά για όλα τα τρόφιμα. Ευχαριστώ. Σα Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Δεκάστρο, τελευταίος μας ομίλητης. Ευχαριστώ συνάδελφε. Ήθελα να προσθέσω κάνα δύο σκέψεις. Η κυρία Κάντεμπαχ κάπως με κάλυψε. Πρέπει να, να μπορεί ο καταναλωτής τελικά να κάνει με επίγνωση επιλογές. Δεν μπορούμε να τον σπρώξουμε μια κατεύθυνση, αλλά με επίγνωση να κάνει την επιλογή του. Το λέω γιατί υπενθυμίστηκε αυτό στο πρώτο πάνελ μέσω άλλων μορφών εκτεθεσίας που επηρεάζονται οι αγορές, όπως αυτά τα, σήματα της τροχέας με κόκκινη ετυχέτα, άμα εμφανίζεται κάτι, δεν είναι κάτι που βοηθάει να κάνει ο καταναλωτής μία επιλογή ε, συνειδητή, αλλά επηρεάζει τη συμπεριφορά του. Τώρα στρεφόμενος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγώ ε, ε, εκτιμώ το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Επίτροπο Ανδρουκάητη έχει κάνει βήματα πρόοδου. Η δουλειά που κάναμε όμως εδώ στο Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή Γεωργίας και στην Ολομέλεια, σε θέματα ετικετοθεσία προέλευση που εφαρμόζεται υποχρεωτικά, είναι κάτι που δεν ελήφθη σχεδόν καθόλου υπόψη. Ο συνάδελφος Ρικ Αντριέ το είπε σαφώ: Θα πρέπει να μπορεί ο καταναλωτή να επιλέγει. Πρέπει να δημιουργήσουμε τι κατάλληλε συνθήκε μέσω πληροφόρηση του καταναλωτού. Από αυτή την έποψη, μεταξύ άλλων, το υπενθύμησε και για το μέλι ο συνάδελφο Χέρντο. Μπορούμε να δώσουμε και άλλα παραδείγματα. Η παραγωγή, α πούμε, κονσέρβα ντομάτα. Οι Ισπανοί, οι Ιταλοί, οι Πορτογάλοι. Πολύ συχνά αντιμετωπίζουν στρέβλους ανταγωνισμού, διότι υπάρχουν κάποιοι παραγωγοί που εισάγουν κινεζικέ ντομάτε και μετά γίνεται πορτογαλική ντομάτα αυτή, η ισπανική ντομάτα. Η ετικετοθεσία προέλευση που εφαρμόζεται υποχρεωτικά θα συμβάλλει στη λύση του προβλήματος. Βέβαια, σε ρυθμιζόμενο επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λαμβάνοντα υπόψη όμως τα πειράματα που κάναμε Εμεί οι οκτώ χώρε που έκαναν αυτό το πείραμα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη με μεγαλύτερη προσοχή αυτό το θέμα μετά θα ήθελα να ζητήσω από την εκπρόσωπο της Food and Drink Europe κάτι. Μίλησε για 45% παραπάνω κόστος για την υποχρεωτική ετικετοθεσία από το ιταλικό πείραμα που κάναμε. Νομίζω ότι αυτό το αριθμητικό στοιχείο είναι κάπως υπερβολικό. Ξέρω, δεν ξέρω τι υπολογισμούς κάνατε. Εγώ το ξέρω, διότι συζητήσεις επανειλημμένα κάναμε στο Κοινοβούλιο αυτό το θέμα. Δεν είναι ένα θέμα που όλοι έχουν ίδια άποψη από αυτού, θα πρέπει όμως να καταλήξουμε σε ένα σημείο σύγκλησης που θα είναι ένα σημείο που θα λαμβάνει υπόψη εκείνο που θέλουν οι καταναλωτές πολίτες. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστούμε συνάδελφοι για τις ε, ερωτήσεις και τα σχόλιά σας. Θα δώσω τώρα το λόγο στους καλεσμένους μας για να σχολιάσουν να θέλουν κάτι, να απαντήσουν σε ερωτήσεις. Ας ξεκινήσουμε ανάποδα. Πρώτα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή. Ευχαριστώ. Να απαντήσω στο σχόλιο που ακούσαμε για το μέλι και την ανάμειξη κινέζικου μελιού με ευρωπαϊκά μέλια. Η αρχή προβλέπει ότι οποιοδήποτε ασφαλέ τρόφιμα μπορεί να τεθεί σε εμπορία στην ευρωπαϊκή αγορά. Και δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε την ε, επισήμανση, την αναφορά της προέλευσης ε, με τρόπο ώστε να χαρακτηριστεί εμπορικό φραγμός. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι χρησιμοποιούμε την υποχρεωτική αναφορά της προέλευσης για να αποτρέψουμε την ε, ε, κυκλοφορία στην αγορά του κινέζικου μέλιου. Από τη στιγμή που το κινέζικο μέλι κρίνεται ασφαλές, ε, έχει θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, από τη στιγμή που χρησιμοποιείται, υπάρχει ανάγκη να ενημερώνουμε κατάλληλα του καταναλωτή, ώστε να γνωρίζει αν το προϊόν που αγοράζει είναι ευρωπαϊκό ή κινέζικο. Και αυτός θα πρέπει να είναι ο στόχος οποιασδήποτε επισήμασης, ε, ε, υποχρέωση επισήμασης της προέλευσης. Ως προς τα σχόλια του κυρίου Αντριέ, δεν θεωρώ ήταν ομή η, η βάναυση, η παρέμβαση του, αλλά άδικη θα τη χαρακτηρίζω εγώ. Ε, αντιλαμβάνομαι την απογοήτευσή σας, ε, γιατί είστε υπέρμαχος της διαφάνειας και προσβλέπετε σε μια θετική έκβαση ε, των πληροφοριών για την προέλευση. Αλλά όταν θέσουμε όλα αυτά στο κατάλληλο πλαίσιο και λάβουμε υπόψη ότι από το 1975 η επισήμανση της προέλευσης ε, θεωρείται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ως ε, εμπόδιο στην εσωτερική αγορά. Μέχρι σήμερα αυτή ήταν παραδοσιακά η νομολογία ε, του ΔΕΚ και η παραδοσιακή θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λόγω του νομικού πλαισίου που μας δεσμεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπετε όμως τι ε, τεράστια πρόοδο είχαμε και νομοθετικά αλλά και πολιτικά τα τελευταία χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχουμε πολύ μεγάλο άνοιγμα πια σε ό,τι αφορά την, τις πληροφορίες για την προέλευση. Έχουμε πραγματοποιήσει ε, επαναστατική θα έλεγα, ρηξικέλευτη πρόοδο τελευταία για το θέμα αυτό. Ήδη είχαμε πρόβλημα με την αντίδραση του Καναδά για την υποχρέωση αυτή. Και παρόλο που σίγουρα υπάρχει επιθυμία να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών, δεν μπορούμε παρά να εφαρμόσουμε την κοινοτική νομοθεσία και να ε, προσπαθούμε να συνδυάσουμε τις διάφορες πτυχές του καταναλωτή, της εσωτερικής αγοράς, των διεθνών μας εμπορικών σχέσεων. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα λοιπόν για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μπορεί εύκολα να θεσπίζει υποχρεωτική αναφορά προέλευσης ε, για τα τρόφιμα. Αλλά ακόμη και όταν ε, δεν είναι υποχρεωτική η αναφορά προέλευσης, ουσιαστικά ενεργοποιείται από την εθελοντική ή υποχρεωτική αναφορά και χρειάστηκε παρόλα αυτά πέντε χρόνια για να εφαρμοστεί. Όχι, μόνο, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ήθελε να θεσπίσει εκτελεστικό κανονισμό, αλλά επειδή ήταν πολύ επίμαχο το θέμα και υπήρχε μεγάλη διάσταση απόψεων. Γιατί θα πρέπει και τα κράτη-μέλη να συμφωνούν και οι δύο συνομοθέτε να εγκρίνουν την πρόταση. Τελικά, όταν προτείνουμε κάτι, φροντίζουμε από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να έχουμε την σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών. Γι' αυτό είναι τόσο χρονοβόρα η διαδικασία. Και δεν έχουμε λάβει ακόμη καμία έκθεση από τα κράτη-μέλη για την εφαρμογή των εθνικών συστημάτων. Περιμένουμε αυτές τις μελέτες, αυτές τις εκθέσεις για να ε, εγκύψουμε διεξοδικά σε αυτές. Ευχαριστώ κύριο Σκαρά. Ευχαριστώ. Να απαντήσω στις διάφορες παρεμβάσεις. Σίγουρα η ανησυχία για τον τομέα υπάρχει. Και πρέπει να πω ότι διαφάνηκε στη συνάντηση που υπενθυμίστηκε πριν, στις 23 Ιανουαρίου νεστότος έτους, στο φόρουμ αυτό που έγινε, στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ για το ρύζι. Εγώ είμαι αισιόδοξο εν γέννη και πρέπει να πω ότι το 2013 είχαμε μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ήταν μειοπική όσον αφορά τα προβλήματα εισαγωγή από τι χώρε με μηδενικού δασμού. Αλλά χάρη στη δουλειά που κάναμε όλοι μαζί, μαζί με τη Γαλλία, μαζί με την Ισπανία και με άλλε χώρε με πολλά άτομα που είναι εδώ παρόντα. Με τα στοιχεία τη ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδείξαμε ότι κάτι δεν λειτουργούσε, δεν πήγαινε καλά όσον αφορά την εισαγωγή με μηδενικό δασμό. Και πρέπει να πω ότι κομβικό σημείο ήταν αυτό το έγγραφο, το Development Solutions. Δηλαδή, όταν ε, πρέπει να γίνει επαλήθευση των συνεπειών, των συμφωνιών αυτών που συνάπτονται με χώρε και αποδεικνύεται ότι για το ρύζι και τη ζάχαρη διαπιστώνονται Σημαντικέ, αξιόλογε ανθρωπιστικές παραβιάσεις και παραβιάσει πολιτικών δικαιωμάτων, αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Δίκαιο έχει και ο Ντόφμαν όταν λέει ότι στην Καμπότζη πιθανότατα η Καμπότζη δεν έχει καν δικαίωμα να θεωρείται μια χώρα που μπορεί να μπει στα everything but arms. Σε αυτές τις χώρες λοιπόν υπάρχουν ευρωπαϊκά συμφέροντα που θέλουν να έχουν εγκαταστάσεις για τη μεταποίηση του ρυζιού το έχουμε επισημάνει εδώ και κάποιους μήνες αυτό στην Όλαφ όταν σε διάφορες ε, τοποθεσίες αμερικανικές υπήρξαν καταγγελίες ενώσεων, παραγωγών ότι, ε, από την Καμπότζη ότι γίνονται τριγωνικά σχήματα. Όλα αυτά πρέπει να προσεχθούν και χρειάζεται επεξεργασία όπως κάναμε μέχρι τώρα και εργασία όπως κάναμε μέχρι τώρα ενωμένοι να κινηθούμε πρέπει να υπάρχει δυνατότητα διαφύλαξης του τομέα, προφύλαξης του τομέα, διότι επαναλαμβάνω. Ένα παράδειγμα κοινού παρανομαστού είναι πώς η οριζοκαλλιέργεια έχει σημασία περιβαλλοντική. Στην Ιταλία, στις, ε, ε, στις εκβολές του Ροδανού, του Πάδου στην Ιταλία, στην Ισπανία, στις εκβολές του Γουαλδικιβίρ, η καλλιέργεια του Ριζιού εμποδίζει ε, στο να μπει το θαλάσσιο νερό στο έδαφος. Οπότε παραμένουν έφορες γέες που δεν θα ήταν έφορες. Αυτό είναι ένα από τα πολλά παραδείγματα που θα μπορούσα να δώσω. Στη συνάντηση της 23ης Ιανουαρίου, πέρα από το θέμα της ρήτρα διαφύλαξης και πέρα από το θέμα της ετικετοθεσίας που δεν έλυσε το δίλημα εθελοντικό υποχρεωτικό το μέτρο, κάτι υπενθυμίστηκε πριν, εκεί υπενθυμίστηκε και το θέμα της αμοιβαιότητας από πλευρά κοινωνικής και περιβαλλοντικής. Κατά την άποψή μας χρειάζεται και μια επανεξέταση του θέματος ε, της ανοχής ε, και θα πρέπει να εξεταστεί και το ενδεχόμενο ενημερωτική εκστρατείας διαφημιστικής πέρα από αυτή που έγινε μέχρι τώρα μέσω του κοινοτικού κανονισμού. Και όσο μας αφορά ε, σε ιταλικό επίπεδο εμάς, πιστεύω πιστεύω ότι έχοντας λύσει κάποια τεχνικά και διοικητικά προβλήματα στη χώρα μας, θα ξεκινήσουμε σύντομα μία εκστρατεία ε, ευαισθητοποίηση όσον αφορά την Ιταλική παραγωγή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γιάκοψ. For... Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ για τις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις σας. Θα προσπαθήσω να τις συνοψίσω στην απάντηση. Κανένα δεν διαφωνεί με το αίτημα για περισσότερη διαφάνεια. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε εδώ. Και είμαστε σαφώς υπέρμαχοι της διαφάνειας. Το πρόβλημα ανακύπτει όταν κάτι τέτοιο οδηγεί σε διαχωρισμό της παραγωγής, σε σπατάλη τροφίμων, σε υψηλότερες τιμές καταναλωτή, σε υψηλότερες ε, τιμές ε, πρώτων υλών και σε μερικές περιπτώσεις δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό βρισκόμαστε σε κάποιο διέξοδο μερικές φορές αυτήν την άποψη. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να εξετάσουμε τα εθνικά μέτρα πιο διεξοδικά και προτείνω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το κάνει αυτό με πιο εναρμονισμένο τρόπο, όχι με 8 διαφορετικές εκθέσεις που με διαφορετικό τρόπο θα υπολογίζουν, θα καταμετρούν τον αντίκτυπο του εμπόριου, στις επιχειρήσεις, στους καταναλωτές και ούτω καθεξής. Είναι σημαντικό επίσης να αναγνωρίσουμε ότι δεν μιλούμε για τη, μόνο την παροχή πληροφορία στον καταναλωτή από τη σκοπιά του επιχειρηματία. Πρόκειται για ένα ολόκληρο σύστημα που θα πρέπει να δούμε αν είναι κατάλληλο με το σκοπό που εξυπηρετεί. Αν υπάρχει συμφέρον του καταναλωτή, ενδιαφέρον του καταναλωτή, ε, επιθυμία για καταβολή της ε, μεγαλύτερη τιμή, ε, τότε σίγουρα αν υπάρχει εμπορικό πλεονέκτημα και οι επιχειρήσει θα είναι πρόθυμε να το κάνουν. Θα πρέπει να βοηθήσουμε του κλάδου που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες. Μιλήσαμε για το κλάδο του ρυζιού, το γαλακτοκομικό κλάδο και σίγουρα η παραγωγή και οι μεταποιητέ ε, είναι αλληλοεξαρτώμενοι. Θα πρέπει να βοηθήσουμε λοιπόν και τους αγρότες αλλά να βρούμε τη σωστή λύση και να προωθήσουμε τα ποιοτικά προϊόντα που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν έχουμε την εσωτερική αυτή συζήτηση απλώ για την εσωτερική αγορά. Η κυρία Κοζουόφσκα. Σας ευχαριστώ. Και εγώ συμφωνώ με τον προλαλήσαντα ότι από τη σκοπιά των επιχειρηματιών πολλά έχουν γίνει και μελέτες της αγοράς και οι επιχειρηματίες φυσικά προσπαθούν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των καταναλωτών. Και πολλές λύσεις έχουν δοθεί και πολλές, πολλές νοτεριστικές λύσεις ε, προκειμένου να ανταποκριθούμε σε αυτά τα αιτήματα των καταναλωτών. Μας ενδιαφέρει φυσικά η γνώμη των καταναλωτών, κυρίως τους επιχειρηματίες, αλλά θα πρέπει οι διατάξεις, οι νομοθετικές διατάξεις που θα θεσπιστούν για τον τομέα αυτό να ε, εφαρμόζεται σε όλους ε, από όλους τους επιχειρηματίες και να μην μπορούν μόνο λίγοι και εκλεκτοί επιχειρηματίες να προσαρμοστούν. Επίσης θα πρέπει να διευκολύνουμε τους επιχειρηματίες να προσαρμοστούν στις αλλαγές, ε, έχοντας σταθμίσει προηγουμένως ε, όλα τα υπέρ και τα κατά των δύο συστημάτων υποχρεωτικής ή εθελοντικής αναφοράς και όλα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη προηγουμένως. Αντί απλώς εθελοντικά ε, να δίνεται η πληροφορία για την προέλευση προκειμένου να ικανοποιηθούν οι καταναλωτές γιατί δεν έχουν όλοι, τη δυνα... όλοι οι επιχειρηματίες τη δυνατότητα να το κάνουν και γι' αυτό είμαστε υπέρ πανευρωπαϊκών λύσεων υπέρ εναρμονισμένων λύσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο έτσι θα έχουμε πρόοδο για όλους ευχαριστώ Μάλιστα, σας ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή στη συζήτηση. Ευχαριστώ τους καλεσμένους. Και τώρα για τα τελικά συμπεράσματα θα ξαναδώσω το λόγο στον πρόεδρο ε, τον κύριο Δεκάστρο. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν συμπεράσματα να συναγάγουμε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους που μίλησαν εκ βάθους καρδίας. Εξετάσαμε από διάφορες γωνίες τις απόψεις που αφορούν το πολύ ευαίσθητο αυτό θέμα, πάρα πολύ σημαντικό θέμα όμως της ετικετοθεσίας προέλευσης των ε, προϊόντων, των τροφίμων εμείς ε, ευχόμεθα η βούληση της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου να μπορέσει σε επόμενες ευκαιρίες ε, να μπορέσει να εφαρμόσει τις ε, προτάσεις, να δώσει υλοποίηση στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είμαστε πεπισμένοι ότι αυτό το θέμα χρειάζεται περαιτέρω εμβάθυνση. Υπάρχουν διάφορες απόψεις, υπάρχουν διάφορες οπτικές γωνίες, που πρέπει να εξεταστούν εις βάθος, οπότε παρόμοιες πρωτοβουλίες με την Επιτροπή Περιβάλλοντος, με την Επιτροπή Γεωργίας από κοινού να το θέμα, μπορούν να ενισχυθούν και να εξεταστούν και άλλες πτυχές εις βάθος και αυτές θα μπορούσαν να βοηθήσουν να θεσπίσουμε νομοθεσία με επίγνωση του θέματος και να βρίσκουμε και σημεία που μπορούν να οδηγήσουν σε βάθυνση της προστασίας των Ευρωπαίων πολιτών και καταναλωτών. Θα σταματήσω, δεν θα προσθέσω κάτι άλλο. Πιστεύω ότι ήταν ένα απόγευμα σημαντικό. Δυστυχώς τη Δευτέρα το απόγευμα και στους φιλοξενούμενούς μας δεν είναι και η καλύτερη μέρα για να διεξάγονται αυτές οι συναντήσεις, διότι οι βουλευτές μας φτάνουν κυρίως Δευτέρα απόγευμα ή βράδυ στις Βρυξέλλες. Δεν είδατε γι' αυτό πολλούς συναδέλφους παρόντες, αλλά Σίγουρα ήταν μια σημαντική ευκαιρία για να κάνουμε βήμα προόδου. Ευχαριστώ όλους και καλό σας βράδυ και καλή επιστροφή.